Okay, colleagues, let's start. Συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε. Καλημέρα, αυτοί οι συνάδελφοι. Σας καλωσορίζω σημερινή συνεδρίαση. Έχετε την ημερήσια διάταξη. Δεν μου είπε κανείς ότι θέλει κάποια αλλαγή. Οπότε περνάμε στο σημείο 2, ανακοινώσει του Πρόεδρου. Εδώ θέλω να αναφέρω πως οι προετοιμασίες για τη διάσκεψη της 14ης Μαρτίου, σε δύο εβδομάδες δηλαδή, με τους προσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων πήγαιναν μια χαρά. Έχουμε ένα πρώτο σχέδιο προγράμματος το οποίο το έχουμε συζητήσει με τον κύριο Μιλητή, τον κύριο Μύρο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ε, Ανοικοδόμησης ε, και Ανάπτυξης και μετά θα υπάρχει ο Φίλιπ Μάιστατ για το δεύτερο κομμάτι, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το βράδυ χάρη στην Περβάνς καταφέραμε να έχουμε τον Ζακ Ντελόρο μιλητή οπωσδήποτε κάτι το πολύ ενδιαφέρον. Ε, δηλώθηκε συμμετοχή από πάνω από 20 κοινοβούλια, μεγάλη παρουσία και έχουμε και απαντήσεις στα ερωτηματολόγια από 15 κοινοβούλια, πάνω από τα μισά. Οπότε Είμαστε μέχρι στιγμή σχετικά ικανοποιημένοι. Αυτά μέχρι τώρα. Ξέρετε πως μετά θα φάμε και ένα δείπνο με την Επιτροπή ε, Οικονομικών Υποθέσεων καθώς τρίτη πρωί 15 Μαρτίου θα συνεδριάσουν και αυτοί με εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Περνάμε τώρα στο σημείο 3, έγκριση των πρακτικών της τελευταία συνεδρίασης, τα οποία έχουν μεταφραστεί και μοιραστεί, δεν ζήτησε κανείς κάποια αλλαγή, οπότε θεωρώ πως εγκρίνονται. Τώρα ερχόμαστε στο βασικό θέμα του σημερινού πρωινού. Το θέμα είναι λοιπόν να δούμε τις μεγάλες αδρές γραμμές της έκθεσης, την δομή της έκθεσης συστάσεις και τα συμπεράσματα. Δεν έχουμε ακόμα την έκθεση δηλαδή, αλλά έχουμε μια λεπτομερή πρόταση για τη δομή της έκθεσης και ποια είναι τα βασικά σημεία που θα αναφέρονται στα κεφάλαια. Αυτό συζητήσουμε σήμερα. και βεβαίως υπερβάνος Θα μας τα βασικά σημεία και μετά θα το συζητήσουμε και ζητώ από όλα τα μέλη και τους ηγητές βεβαίως να τοποθετηθούν. Περιμάνος, έχεις τον λόγο. Euh, euh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή στη σχέση με την τελική εργασία της ε, ομάδας ε, εργασίας μας γιατί βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη δεύτερη φάση των εργασιών διαπιστώνω ότι διαφοροποιηθήκαμε σε σχέση με το πρώτο τμήμα της ε, άσκησής μας. Στο τμήμα, στη διάρκεια του πρώτου του τμήματος είχαμε την δυνατότητα να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων επί της ουσίας μεταξύ μας και νομίζω ότι όλοι επιθυμούν αυτό το τελευταίο κομμάτι της Επιτροπής Κρίσης ε, να λάβει χώρα με πιο ήρεμο τρόπο. Εξού και η πρόταση για τη σημερινή συνεδρίαση πριν καν να αρχίσω τη συγγραφή του οριστικού σχεδίου έκθεσης. Σκέφτηκα ότι μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας μπορεί να αποσαφηνίσει τους ακατάρθους στόχους, γιατί η προσπάθειά μας θα είναι συλλογική. Και μάλιστα, όταν θυμάμαι τις ανταλλαγές επί που είχαμε, πέραν ε, των ανταλλαγών απόψεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια και την, Εθνική, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώνω ότι μέχρι στιγμής είχαμε μεταξύ μας μία συζήτηση προς ανατολισμού. Κατά το δεύτερο τμήμα των εργασιών μας. Και αυτό που χαράχθηκε στη μνήμη μου ως κατακλείδα αυτών των ανταλλαγών απόψεων και ιδιαίτερα κάποιες παρατηρήσεις του Φρανκ Ράγκελ και δικέ σας κύριε Πρόεδρε. Αυτό που μου έμεινε λοιπόν είναι το εξής. Καταρχήν όλα τα κεκτημένα από την πρώτη έκθεση θα πρέπει να παραμείνουν ως κεκτημένα. Δεν χρειάζεται να ξανανοίξουμε για αυτά τη συζήτηση. Με τον Ότμαρ Κάρας είχαμε συζητήσει και το θέμα αν θα, πρέπει να περιοριστούμε στο να θέσουμε κάποιες ερωτήσεις ή θα μπορούσαμε να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι και να θέσουμε κάποια στρατηγικά ζητήματα ε, για το μέλλον. Και χάρη στην ε, συνεργασία και την πολιτική βούληση των μελών της Επιτροπής επιλέξαμε τη δεύτερη εναλλακτική λύση και η ενδιάμεση αυτή έκθεση περιλαμβάνει πολύ σημαντικά συμπεράσματα ως προς την ουσία για τον προσανατολισμό και το ευρωπαϊκό μήνυμα που θέλουμε να προκύψει από τις εργασίες της Επιτροπής μας. Δεν προτείνω λοιπόν να ξανασυζητήσουμε τα σημεία της πρώτης έκθεσης. Και μάλιστα αυτό το κανόνα θα ακολουθήσω και κατά την κατάρτιση της δεύτερης έκθεσης. Το δεύτερο σημείο που είναι σημαντικό επίσης είναι ότι όπως και κάτι, κατά την πρώτη περίοδο της εντολής μας προσπαθήσαμε να μείνουμε ως προς το έργο των υπόλοιπων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Δηλαδή όλο το πακέτο της οικονομικής διακυβέρνησης που αποτελεί αρμοδιότητα της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το μηχανισμό κυρώσεων ή την ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας. Όλα αυτά τα θέματα που είναι αρμοδιότητα άλλων επιτροπών δεν πρόκειται να απασχολήσουν και εμάς. Δεν πρόκειται να ασφετεριστούμε αρμοδιότητες άλλων επιτροπών. Φυσικά όλα αυτά τα σημεία είναι σημαντικά και για μας και για όλους φυσικά. Αν όμως μέσω αυτής της τελικής μας έκθεσης προσπαθέσουμε με μη νομοθετικό τρόπο να πούμε κάτι που αλλού λέγεται με νομοθετικό τρόπο, δεν νομίζω ότι ε, χρησιμοποιούμε με το βέλτιστο τρόπο αξιοποιούμε στο έπακρο το περιεχόμενο αυτής της τελικής έκθεσης. Και δεν θα πρέπει σε αυτή την τελική έκθεση να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε κάποια σημεία από τα οποία μείναμε δυσαρεστημένοι από το νομοθετικό πακέτο. Επίσης, ε, θα ήθελα να πω ότι στην συζήτηση προσανατολισμού που είχαμε στις αρχές της ανανέωσης της εντολής μας καταλήξαμε και σε ένα άλλο συμπέρασμα. Να εξετάσουμε με φιλόδοξο τρόπο και με μια ευρωπαϊκή προσέγγιση που είναι κοινή για την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής μας και να υιοθετήσουμε μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική. Νομίζω ότι μεταξύ μας είχαμε συμφωνήσει. Βέβαια κάποιοι διαφωνούν, <coughs> ας το δηλώσουν. Αλλά νομίζω ότι είχαμε μεταξύ μας συνεννοηθεί ότι επευκαιρία αυτή αυτής της έκθεσης Επιτροπής για την κρίση καλό θα ήταν να εξετάσουμε το πώς είναι σκόπιμο να εξελιχθεί στο μέλλον το κοινοτικό δίκαιο για να ανταποκριθούμε στο ύψος των φιλοδοξιών μας. Και αν σήμερα έχουμε δεσμευτεί για μία αναθεώρηση της συνθήκης που σχετίζεται με τη συγκυρία της διαχείρισης του δημόσιου χρέους, πολλοί πιστεύουμε ότι δεν είναι αυτή η τελική αναθεώρηση της συνθήκης και θα πρέπει να έχουμε και μια ενδιάμεση αναθεώρηση ή να θεσπίσουμε μια ενισχυμένη συνεργασία στην Ευρωζώνη. Και ότι αυτή η έκθεση θα έπρεπε να μας δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα για τη συζήτηση αυτή. Και ελπίζω να επιβεβαιώσετε το γενικό αυτό προσανατολισμό. Επανέρχομαι λοιπόν στο έγγραφο. Δεν θέλω να επαναλάβουμε συζητήσεις του παρελθόντος και κυρίως να αποφύγουμε μια παρεκτροπή της συζήτησης ή υπερβολική περιπλοκή. Γιατί έτσι θα χαθούμε και θα πελαγοδρομήσουμε. Ελπίζω κατά το τέλος της συνεδρίασης να έχουμε μία επιβεβαίωση ως προς την διάρθρωση και τη δομή της έκθεσης. Δεν θα ήθελα να εμπλακούμε σε μια βυζαντινολογία και να καταλήξουμε σε πολύ γενικά και όριστα συμπεράσματα ως προς τη δομή της έκθεσης. Εγώ απλώς σας προτείνω να επανέλθουμε στις έξι βασικές ερωτήσεις που ομόφωνα ενέκριναν και οι συντονιστές. Γιατί με την ανανέωση της ε, θητείας μας, της εντολής μας, καθορίσαμε έξι ζητήματα γύρω από τα οποία οργανώσαμε τις δημόσιες ακροάσεις μας, γύρω από τις οποίες οι πολιτικές ομάδες ε, οργάνωσαν τις ε, συνεδριάσεις τους. Και δεν θα ήθελα να απομακρυνθούμε από αυτά τα σημεία. Αν θέλετε να μιλήσουμε για τη δομή, να το κάνουμε αλλά να μην αμφισβητήσουμε αυτά που είχαμε αποφασίσει στην αρχή της ανανέωσης της εντολής μας. Δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο προς το τέλος της εντολής να αμφισβητήσουμε αυτά που είχαμε αποφασίσει στην αρχή της. Επίσης, στη δεύτερη φάση αυτού του εγχειρήματο, στη δεύτερη φάση της εντολής, είχαμε αποφασίσει να έχουμε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Θέλουμε στο έργο μας να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της διακυβερνητικής μεθόδου και της κοινοτική με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει τεράστια εμπειρογνωμοσύνη. Αυτό είχαμε αποφασίσει και επιδιώξει. Και επίσης είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε συζήτηση με τα εθνικά κοινοβούλια. Μερικές φορές οι συνθήκες ήταν αντίξωες γιατί το πρόγραμμά μας ήταν φορτωμένο, κάτι που περιέπλεξε τη διοργάνωση των επαφών, αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι αξιοπρεπέστατο γιατί είχαμε συνεδρίαση με εκπροσώπους της Ολλανδικής και της Γαλλικής Βουλής και επίσης είχαμε μια πολύ επιτυχημένη αποστολή στην Πορτογαλία, κάπως πιο περίπλοκη στην Ισπανία. Δύο πολύ σημαντικές χώρες υπό το πρίσμα της αξιολόγησης της κρίσης που θα κάνουμε σήμερα. Είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων και στη Γερμανία, θα στείλουμε αποστολή και στην Ελλάδα. Είχαμε μια πληρέστατη αποστολή στο Ηνωμένο Βασίλειο και μια σύντομη ανταλλαγή αλαμεστή στην Τσεχία. Άλλωστε, όπως είπατε, 15 εθνικά κοινοβούλια ήδη απάντησαν στις 7 ερωτήσεις που τους είχαμε στείλει. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε τώρα στο κυρίω θέμα, τα έξι θέματα που θα αποτελέσουν τους άξονες της τελικής μας έκθεσης έξι αυτά τα θέματα φυσικά περιστρέφονται γύρω από το ζήτημα του δημόσιου χρέους και της κρίσης του ευρώ. Και θα πρέπει να μην μείνουμε εγκλωβισμένοι στις μέχρι τώρα συζητήσεις ε, της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής για τα έξι νομοθετικά κείμενα, αλλά να είμαστε και λίγο πιο φιλόδοξοι για να δούμε πώς θα δημιουργήσουμε ένα πραγματικό Ευρωπαϊκό Υπουργείο Οικονομικών κατά κάποιο τρόπο και αν πέραν του μηχανισμού που προβλέπει η συνθήκη μπορούμε να δούμε ένα, πώς, ε, ένα ζήτημα κοινή αντιμετώπισης του χρέους όπως πρότειναν ο κύριος Τελπλά ή άλλοι για ένα ποσοστό τουλάχιστον του δημόσιου χρέους ε, που θα αντιμετωπιζόταν από κοινό τρόπο. Το δεύτερο ζήτημα όσον αφορά λοιπόν τις ε, παγκόσμιες ανισορροπίες ε, και την συνολική διακυβέρνηση, εδώ πιστεύω ότι εμπίπτουν τρία ζητήματα, τα οποία χρήζουν περαιτέρω ανάπτυξης. Το πρώτο αφορά την ε, ισορροπία που διαφαίνεται ήδη στην ενδιάμεση έκθεση και η οποία σιγά σιγά προχωράει. Δηλαδή τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο και χαίρομαι που ε, η νέα πρόταση, ε, κατά κάποιο τρόπο δηλαδή μου δίνει τη δυνατότητα να έχω μια σύνοψη πριν από την τελική σύνοψη και χαίρομαι που αναφέρεται αυτό, αυτή η ανησυχία ε, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ε, μπορούμε να βγάλουμε την Κίνα από τις πολυμερείς ε, συμφωνίες από τη στιγμή που αυτό κινδυνεύει τελικά να γίνει σε διάλογος ανάμεσα στην Κίνα και τη ΣΥΠΑ. Το δεύτερο ζήτημα, το οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει εδώ, είναι το ζήτημα της πρόσβασης ε, στις πρώτες ε, ύλες. Η λειτουργία λοιπόν της αγοράς ε, πρώτων υλών γιατί ξέρουμε ότι ο ΖΕ20 θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό αλλά ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να αναπτύξουμε και το θέμα αυτό. Τρίτο σημείο αφορά γενικότερα την λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Επ' αυτού διαπιστώνουμε σειρά κακών πρακτικών. αζοπυρώθηκαν με πολλές κακές επιπτώσεις για την πραγματική οικονομία και θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας. Εδώ, στην έκθεσή μου, αναφέρω ε, σαφώς ε, την, ε, την συνένωση της Deutsche Börse και της Nice Euronext που αφορά την συνέχεια, ενδεχομένως όχι το τέλος, αλλά πάντως τη συνέχεια μιας σειράς επεισοδίων που καταδεικνύει, εν πάση περιπτώσει, την ε, ισχύ κάποιων πρωταγωνιστών της ε, ε, οικονομίας και αναφέρομαι εδώ γενικότερα στις μεγάλες επενδυτικές τράπεζες που ξέρουμε ότι χειρίζεται τα κεφαλαία του η Deutsche Börse. Το ζήτημα αυτό έπρεπε να βρίσκεται στην έκθεσή μας γιατί δεν αναφέρεται πουθενά στα νομοθετικά κείμενα τα οποία φτάνουν ε, σε μας. Ε, ε, βεβαίως στην έκθεση της ε, Επιτροπής ε, Νομισματικών Υποθέσεων οπωσδήποτε θα υπάρχει σε ένα δεύτερο πίσω πλάνο σαν υπόβαθρο γενικότερη οικονομική κατάσταση αλλά πιστεύω ότι πρέπει να αναφερθεί σαφέστερα. Και από την άλλη πλευρά εδώ ε, ε, πρέπει να ρωτήσουμε, να αναρωτηθούμε τι σημαίνει και μια πραγματική εποπτεία για τέτοιους πρωταγωνιστές της αγοράς. Και από την άλλη πλευρά ποια είναι η συμβολή τέτοιων οργανισμών στην πραγματική οικονομία. Γιατί ένα από τα μηνύματα κλειδιά και της πρώτης έκθεσης και που βρίσκεται και αλλού και το λέω, το αναφέρουμε συνέχεια, είναι ότι αυτοί οι οργανισμοί θα πρέπει να συμβάλλουν στην χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Αλλά αυτού του είδους οι συγχωνεύσεις εγκυμονεί τον ε, σημαντικό κίνδυνο της, ε, ε, του να έχουν την οικονομία στα χέρια τους ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και η οικονομία να βασίζεται σε αυτές τις χρηματοπιστωτικές κινήσεις. ο κίνδυνος ανάπτυξης νέων κερδοσκοπικών φουσκών, ε, κυρίως ε, στην ε, κυρίως στην οικοδομή, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια τέτοια κίνηση, μπορεί να αποβεί εξαιρετικά επικίνδυνη για την οικονομία. Και από την άλλη πλευρά, για την πραγματική οικονομία, η εξαγορά από τρίτα κεφάλαια μεγάλων τμήματων της βιομηχανίας μας. Και αυτός είναι ένας εξαιρετικά μεγάλος κίνδυνος. Και ξέρω ότι ο φίλος Βόλι Σμιτ ε, αμέσω αρχίζει να διαμαρτύρεται λέγοντας ότι ε, είμαι υπέρ του προστατευτισμού. Εγώ πιστεύω πάντω, ότι πρέπει να γίνει η συζήτηση αυτή και να δούμε τα στοιχεία αυτά. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα προχωρήσουμε. Λέμε, ωραία, συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε την πραγματική οικονομία ότι θα πρέπει να δώσουμε προστιθέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, αλλά ενθυμούμενη και στοιχεία του παρελθόντος θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Και για να ολοκληρώσω επί του σημείου αυτού, πρέπει να πω ότι οι μηχανισμοί εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών, έτσι όπως τους έχουμε ε, ορίσει μέχρι τώρα, αφορούν μονάχα την ε, χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Και η Κεντρική Τράπεζα έχει πλέον και μία εντολή όσον αφορά την εποπτεία μακροοικονομικών κινδύνων, αλλά πρόκειται για μία εποπτεία η οποία συνδέεται με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και όχι με τα υπόλοιπα. Δεν συνδέεται δηλαδή ε, με τον τρόπο με τον οποίο τελικά θα χρηματοδοτηθεί η παγκόσμια οικονομία και στην χρηματοδότηση της ε, συγγνώμη, πραγματικής οικονομίας ε, το ζήτημα της διαχείρισης του βιομηχανικού κεφαλαίου είναι πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Επόμενο. Θέλουμε ένα νέο διεθνές νομισματικό σύστημα. Εδώ δεν θα πλατιάσω γιατί πολλής λόγος έχει γίνει ε, για αυτό το ζήτημα και πιστεύω ότι υπάρχει μια συνένεση κατά την οποία ε, ή σύμφωνα με την οποία ε, το, το G20 θα πρέπει να θεσμοθετήσει κάτι τέτοιο, να το συνδέσει με, τη, με τους οργανισμούς Bretton Woods. Η συζήτηση δεν έχει ολοκληρωθεί, ενδεχομένως θα πρέπει βεβαίως να δούμε και μεταξύ μας να συζητήσουμε εάν το σύστημα Bretton Woods θέλουμε τελικά να διασυνδεθεί με την συνολική διακυβέρνηση ανεξάρτητα από τις παγκόσμιες αγορές και εγώ πιστεύω ότι ναι και ότι ε, η Επιτροπή μας έχει την ίδια ε, προσέγγιση. Επόμενο σημείο, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της αηφορίας μέσα στα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια το, του, ε, της στρατηγικής 2020, ανάπτυξη. Και εδώ θα είμαι λακωνική, γιατί ήδη μίλησα πάρα πολύ. Εδώ θα μπορούσαμε να επιμείνουμε επί δύο σημείων. Το πρώτο αφορά την εσωτερική αγορά. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε ήδη στο πρώτο σκέλος της εργασίας μας επ' αυτού στην Επιτροπή ΙΜΚΟ, ΕΚΟΝ, ε, ε, απασχόλησης. Όλοι μελετούν την Single Market Act. Ε, γι' αυτό λοιπόν εγώ προτείνω να μην ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό εδώ σε εμά, να μην το ξανανοίξουμε το κεφάλαιο αυτό, να δούμε βεβαίως τη δυναμική που κρύβεται πίσω από την ενιαία αγορά και να δούμε τη διασύνδεση η οποία υπάρχει μεταξύ της ενιαίας αγοράς και το άλλο πολύ σημαντικό πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δηλαδή αυτή η ιδέα που ακόμα βρίσκεται σε ε, πρωτόλιο στάδιο, δηλαδή να ξεκινήσει μια να ιδρυθεί μια ευρωπαϊκή κοινότητα ενέργειας. Θα ήθελα εδώ να ασχοληθώ με το θέμα της ε, εκπαίδευσης. Πολλά έχουμε πει για το θέμα αυτό, αλλά στην γενικότερη ευρωπαϊκή πρόκληση το ζήτημα της εκπαίδευσης είναι ας πούμε πρόκληση με κεφαλαίο π, αλλά θα μου πείτε υπάρχουν ένα σωρό προκλήσεις τέτοιου είδους. Ε, ε, ε, και στη στρατηγική 2020 και στη Λισαβόνα λέγαμε πώς θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο έτσι ώστε να μην να ξεφύγει από την ένδια, τι πρέπει να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι το θέμα της εκπαίδευσης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Πέμπτο θα πρέπει να ξανασκεφτούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση πέρα από την ε, ε, ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. Είναι αυτά τα οποία αναφέραμε και όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση για την ε, μεταρρύθμιση της συνθήκης και νομίζω ότι όλοι συμφωνούν. Στην Οικονομική Επιτροπή ο Στάνφος Σογιών Λάινεν κατέθεσε τροπολογία για την έκθεση Σουκουλούνα έτσι ώστε να υπάρχει μια δυνατότητα επανέναρξης ε, ε, μελλοντικής μεταρρύθμισης ε, της συνθήκης και προτείνω το περιεχόμενο να μετατεθεί εδώ γιατί είμαι απολύτως πεπισμένη ότι δεν δεν θα μείνουμε εδώ. Ή θα υπάρξει αναθεώρηση της συνθήκης ή θα υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία της Ευρωζώνης. Και σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να είμαστε στην ίδια κατάσταση που είμαστε σήμερα. Σήμερα έχουμε αναθεώρηση της συνθήκης που για πρώτη φορά δεν συνδέει παρά μερικά ε, ή τυπικά μονάχα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δέστε λίγο την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι αναθεωρήσεις και ενισχυμένες συνεργασίες έχουν παραδοσιακά προετοιμαστεί από μια πραγματική πρωτοβουλία η όθηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και βεβαίως δεν αναφέρουμε ούτε στις εκθέσεις Νταφ, ούτε σε άλλες Μπροκ, Μέντες, Δεβίγο, ένα σωρό. Σπινέλη, όσο πιο πίσω πηγαίνουμε βρίσκουμε κι άλλες στοιχεία τα οποία τελικά τροφοδότησαν τις αναθεωρήσεις των συνθήκων. Και εδώ έχουμε το παράδοξο. Για πρώτη φορά το Κοινοβούλιο να έχει επισήμως ε, αρμοδιότητες ε, και τότε δεν γίνεται τίποτα. Και τη στιγμή που ζητάει η αναθεώρηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που αφορά τελικά ε, το αναθεώρηση του τρόπου ψηφοφορίας. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι σημαντικό. Αλλά εάν κάνουμε μια τέτοια κίνηση για να ζητήσουμε αλλαγή του τρόπου εκλογής στις ευρωπαϊκές εκλογές, μπορούμε να το κάνουμε και για άλλα σημαντικά ζητήματα. Ε, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, πολύ σημαντικό ζήτημα. Το λέω και υπό την αίρεση του ελέγχου των συναδέλφων. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό. Εγώ βεβαίως δεν θέλω να ξανανοίξω ε, το θέμα ε, της ε, φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών γιατί τα έχουμε συζητήσει και τα έχουμε ξανασυζητήσει και τα είπαμε και στην πρώτη έκθεση. bientôt le rapport Podimata qui euh, largement euh, euh, porte sur cette question. Ε, ε, αλλά όσον αφορά αυτά τα ομόλογα έργων, τα project bonds, ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, κάνουμε λόγο και για αυτά γιατί είναι και αυτά πολύ σημαντικά. Αυτά ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω τίποτε άλλο και νομίζω ότι έτσι τροφοδοτείται σωστά η συζήτηση. Ευχαριστώ Περβάνς. Τώρα θα ζητήσω να μιλήσουν οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Πρώτα απ' όλα Μπάστος, κατόπιν ο Ρόμπερτ Γκέμπελς, ο Όλε Σμιτ, ο κύριος Χουντής και ο κύριος Μποργέζιο. Α, έφυγε. Οπότε ξεκινάει η συζήτηση για τους υπολείπους. Ο κύριος Μπάστος λοιπόν. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτική και όσο πιο συγκεκριμένη γίνεται. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Μπέρες για τις επεξηγήσεις που μας έδωσε και να πω ότι υπάρχουν δύο διαμετρικά αντίθετες προσεγγίσεις. Η μία η προσέγγιση που μας παρουσίασε εδώ προφορικά η κυρία Μπέρες για το έργο της τελικής έκθεσης που υστερεί σε σχέση με τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό θα αναλύσω αυτά που θεωρούμε ότι είναι αποδεκτά και αυτά που απάδουν από το κείμενο που είχαμε λάβει. Συμφωνούμε με τις έξι ερωτήσεις και τη δομή της έκθεσης. Συμφωνούμε με τη φιλοδοξία της έκθεσης. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση επίσης για την πρόταση να μην επαναλάβουμε τη συζήτηση για τα διάφορα ζητήματα της ενδιάμεσης έκθεσης. Ούτε έχουμε καμία αξίωση ή διεκδίκηση για επικάλυψη του νομοθετικού έργου άλλων καθήλια αρμόδιων επιτροπών. Ως προς αυτά συμφωνούμε απόλυτα με την κυρία Μπέρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στο έγγραφο που μας μοιράστηκε. Πρόκειται για ένα σχέδιο έκθεσης καταρχή που κατά τη γνώμη μας δεν αντικατοπτρίζει, επουδενή, ούτε το περιεχόμενο των συζητήσεων που είχαμε, ούτε την ανταλλαγή απόψεων στα διάφορα εθνικά κοινοβούλια. Γι' αυτό θεωρώ ότι στερεί σε σχέση με τις προσδοκίες μας. Γιατί ούτε είναι τολμηρό το έγγραφο, ούτε διορατικό ή οραματικό προς το μέλλον. Το ΕΛΚ πρότεινε κάποιες θέσεις για την τελική έκθεση, κάποιες παρατηρήσεις. Δεν υπάρχει τίποτα καινούριο ή μερικές φορές αυτές οι θέσεις του ΕΛΚ δεν περιλήφθηκαν καν στις ε, αδερές γραμμές της τελικής έκθεσης. Θα ήθελα να πω ότι το έργο που επιτελέσαμε στην Επιτροπή μας τις τελευταίες εβδομάδες και οι προτάσεις των πολιτικών ομάδων θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση του σχεδίου που θα υποβάλει η γραμματεία ώστε να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε σε αυτά που μας παρουσίασε σήμερα προφορικά η συγγήτρια. Και θα θέλαμε στο έργο αυτό που θα γίνει, τη σύνοψη των προτάσεων των πολιτικών ομάδων, να προσδιοριστούν οι παρατηρήσεις των πολιτικών ομάδων και μάλιστα αναφέροντας ονομαστικά τους εμπνευστές αυτών των ε, προτάσεων και πρωτοβουλίων. Έσω ένα ερώτημα. Μπορείτε λίγο να καθορίσετε. Δουλεύει. μου, θα τα πω αγγλικά. Ακούτε, ακούτε διερμηνία. Λοιπόν, θα τα πω στα αγγλικά. Μπορείτε να μας πείτε ποια, ποια είναι τα σημεία που νομίζετε ότι λείπουν. Κατάλαβα. Νομίζω ότι ήταν ε, φω φανάρι αυτά που είπα, σαφέστατα. είπα ότι οι εξηγήσει που μας έδωσε η κυρία Μπέρες, οι προφορικές εξηγήσει που μας έδωσε σήμερα, περιορίζονται στα συνενετικά σημεία. Δηλαδή, δεν θέλουμε να επαναλάβουμε ή να σφετεριστούμε το έργο άλλων επιτροπών που είναι καθήλυν αρμόδιες. θέλουμε μια φιλόδοξη έκθεση στραμμένη προς το μέλλον συμφωνούμε με τις έξι ερωτήσεις, αλλά το σχέδιο που επίσημα μας υπευλήθη δεν αντανακλά αυτά που ακούσαμε σήμερα προφορικά από την ε, Περβάς Μπέρες. Το σχέδιο έκθεση είναι που απάδει από αυτά που ακούσαμε από την κυρία ε, Μπέρες. Γι' αυτό και ζητήσαμε από την εισηγήτρια και από τη γραμματεία να συντάξουν ένα έγγραφο εργασίας που θα αντικατοπτρίζει αυτά που έχουμε ακούσει πριν από λίγο από την εισηγήτρια και που δεν ε, ε, αντιστοιχούν σε αυτά που έχουμε στο κείμενο. Γιατί με αυτά που είπε η εισηγήτρια πριν από λίγο συμφωνούμε. Αλλά το κείμενο που λάβαμε δεν συμφωνεί με αυτά. Υπάρχει μια αντιστοιχία, υπάρχει μια σαφή αντίφαση μεταξύ αυτών που ακούσαμε πριν από λίγο προφορικά από την εισηγήτρια Μπέρες και του περιεχομένου του σχεδίου έκθεσης. Συνεχίζουμε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ θερμά την Περβάνς για το έργο που έχει επιτελέσει και τη συγχαίρω όχι μόνο γιατί είμαστε στην ίδια πολιτική ομάδα αίματος αλλά γιατί πραγματικά οι προτάσεις της ε, είναι πολύ εμπνευσμένες. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια της κυρίας Μπάστος. Αν κατάλαβα καλά, ζήτησε από τη γραμματεία να υποκαταστήσει τους ευρωβουλευτές στο έργο τους και να προσθέσει γραμματεία αυτά που λείπουν από το, την έκθεση της κυρίας Μπερές. Αυτό κατάλαβα από την παρένεση της κυρίας Μπάστος. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το νόημα μια έκθεση. Η υπερβάστη υποβάλλει την έκθεσή της και οι βουλευτέ θα έχουν ε, το χρόνο να υποβάλουν τροπολογίες και ενδεχομένω να συμπληρώσουν τα κενά που θα διαπιστώσουν ότι παρουσιάζει η έκθεση. Πάντως συμφωνώ με την εισηγητριά μας ότι θα πρέπει να αποφύγουμε να έχουμε επικάλυψη με το έργο των νομοθετικών επιτροπών, γιατί η δική μας επιτροπή είναι επιτροπή προβληματισμού και όχι επιτροπή με νομοθετική αρμοδιότητα. Θα πρέπει να μείνουμε λοιπόν σε αυτό το επίπεδο του προβληματισμού και της εξέτασης. Βέβαια είναι αδύνατο να αποφύγουμε θέματα όπως η οικονομική διακυβέρνηση ή το θέμα των ευρωμολόγων και άλλα παρόμοια. Πάντως θα πρέπει να κάνουμε πάνω δυνατόν ώστε να παραμείνει συνοπτική έκθεσή μας, γιατί αν ε, θέλουμε πραγματικά να μας διαβάσουν, να διαβάσουν την έκθεσή μας και να μας καταλάβουν, δεν θα πρέπει να μετατραπεί σε μια νέα βίβλο η έκθεσή μας, θα πρέπει να περιοριστούμε στα ουσιώδη, να είναι ευσύνοπτη και ευανάγνωστη η έκθεση αυτή. Και θα πρέπει από κοινού να καταδικάσουμε και να στυλιτεύσουμε όλες ε, αυτές οι παρεκτροπές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της παγκοσμιοποίησης. Είναι κάτι κεκτημένο που θα συνεχιστεί, αλλά σίγουρα διαπιστώνουμε κάποια έκτροπα, κάποιες παρεκκλήσεις, όχι μόνο εμάς αλλά και αλλού και θα πρέπει αυτές να τις ε, κατονομάσουμε. Και αυτή είναι η αποστολή μας, να προτείνουμε και κάποιες λύσεις μέσω και μακροπρόθεσμα. Κάποιες λύσεις που θα τις χαρακτήριζα ακόμη και ριζοσπαστικές με την καλή έννοια του όρου. Δηλαδή καινοτόμε, αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστικές. Και φυσικά διαφυλάσσοντας αυτό το όραμα, το όνειρο που είναι απαραίτητο στην πολιτική. Ευχαριστώ, Ρόμπερτ. Περνάμε τώρα στον Σμιτ, όλοι Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Εμείς έχουμε μια παροιμία που λέει πως ε, καμιά φορά το μέλλον μπορεί να σε ευνηδιάσει από πίσω. Ίσως βεβαίως το μέλλον να έχει ήδη φτάσει. Εν πάση περιπτώσει εγώ δεν θεωρώ πως πρέπει να επαναλαμβάνουμε τα πάντα, αλλά υπάρχει μια διαφορετική κατάσταση. Η ιστορία υπάρχει. Ε, και δεν νομίζω πως είναι σωστό να μην αναφέρουμε τα της Βορειοαφρικής και της Μεσανατολής. Εσείς λέτε όχι, εντάξει, μα είναι ουσιαστικό για αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Και νομίζω πως όλοι μας, δεν τουλάχιστον εγώ, είμαι απογοητευμένος από την ευρωπαϊκή αντίδραση αυτό σχετίζεται, ε, αυτά που αναφέρονται στο κείμενο, ε, θεωρώ πως πρέπει να επαναλάβουμε τα πάντα, αλλά κάποιες σκέψεις. Δεν νομίζω πως η κυρία Μπερές θα συμφωνούσε. γιατί τα λέω αυτά. Γιατί έχουμε κάνει έξι σελίδες σχόλια και ένα επιχείρημα ε, εδώ πέρα αναφέρει την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Αναφέρθηκε και στην πρώτη έκθεση. Και βεβαίω αυτό σχετίζεται άμεσα με τα προβλήματα που έχουμε στην Ευρώπη σήμερα. Και κάποιος είπε πως ε, είναι καλύτερο να έχουμε προϊόντα από τη Βόρεια Αφρική από πρόσφυγες. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική μας όσον αφορά το εμπόριο και όσον αφορά την κοινή πολιτική. Δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε τώρα αυτό. Αλλιώς θα είμαστε τόσο κακοί όσο ήμασταν τις τελευταίες δύο-τρεις εβδομάδες. Γιατί, Ρομπέρ, δεν νομίζω πως μπορούμε σε οποιαδήποτε έγγραφα πολιτικής να μην αναφέρουμε το τι συμβαίνει στην επικαιρότητα τους, δεν είναι πολιτισμός. Κάποια σύντομα σχόλια τώρα νομίζω πως θα πρέπει να αναφέρουμε περισσότερο, να μιλήσουμε για κρίση της Ευρωζώνης και όχι ευρωπαϊκή κρίση. Γιατί αν θέλουμε και άλλες χώρες να μπουν στην, ε, στο ευρώ, να πούμε πως δεν είναι πρόβλημα του νομίσματος το πρώτο θέμα αυτό για τα, το δημόσιο χρέος και την κρίση του ευρώ και τα ευρωομόλογα. Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση με την Κομισιόν και τα σχόλια εδώ που έγιναν δεν θυμάμαι από ποιον Μπέριγκαν, από τον κύριο Μπέριγκαν είναι πολύ επιφυλακτικός ε, στο τέλος και αυτό πρέπει να, να φανεί νομίζω. Ξέρω πως υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και εντός της ομάδας μου, αλλά πάντα διαφέρουν οι απόψεις εντός της ομάδας μου. Αλλά νομίζω πως πρέπει, πρέπει να αντικατοπτριστεί αυτό. Πως πρέπει να ξέρουμε εμείς που χαράζουμε πολιτική τι κάνουμε. Και... Ε, να το σκεφτούμε περισσότερο. Τώρα μιλάτε ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Υπουργείο ναι. Οικονομικών, τι εννοείται. Αυτό εννοείται. Ξέρω πως ο πρόεδρος εδώ πέρα θα ήθελε να εξηγήσετε αυτό το, το ταμείο, την παρατήρηση για το γερμανικό χρηματιστήριο και τη της κτλ. Υόρκης και Οπότε το, το αφήνω αυτό. Κατόπιν μεταναστευτική πολιτική και μετά υπαριθμόν 3 ένα νέο νομισματικό σύστημα. Ναι, συμφωνούμε με αρκετά από αυτά, αλλά είναι πολύ εκτεταμένα, ειδικά όσον αφορά τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις. είναι φυκτά αυτά τα πράγματα. Εδώ δεν μπορούμε να λύσουμε τα δικά μας προβλήματα στην Ευρώπη και ζητάμε από τον κόσμο να, να λύσουν όλα τα προβλήματα ζητάτε ένα νέο οικονομικό συμβούλιο ασφαλείας στους G20. Δεν ξέρω, είμαι πολύ επιφυλακτικός. Βλέπετε πώς λειτουργεί και σήμερα το, το Συμβούλιο. Το 4... Εν ολίγης μπορούμε να πούμε περισσότερο ο Μόντι, ότι θέμε. Τρία μη δηλαδή, περισσότερο Μάριο Μόντι. Τρία μη στα αγγλικά βεβαίω. Είναι και μια μάρκα σοκολάτας εκεί πέρα. Υπάρχουν, ναι. Το υπαριθμόν 5, ο φόρος ε, των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Ψηφίζουμε την ερχόμενη εβδομάδα στο Τρασβούργο και η κυρία Ποδηματά έχει κάνει καλή δουλειά εδώ πέρα για να μην πω πως ήταν αδύνατη η αποστολή της, αλλά δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα βεβαίως που θα προκύψει. Βεβαίω, εντάξει. Θα, θα πρέπει να, να υπάρχει μέσα, να, να, λέμε και το τι ψηφίζουμε την άλλη εβδομάδα. Και, και το αποτέλεσμα ίσως να μπει. Το υπαριθμόν 6 να το αφήσω στον, στον πρόεδρο να το δει. Ο κύριος Κλίντς έχει πολλά να πει για αυτά τα ταμεία και το πώς χρησιμοποιούνται. Εγώ θεωρώ πως θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με πιο πρακτικό τρόπο και να στραφούμε περισσότερο σε πιο πραγματική αξία για την Ευρώπη, έργα υποδομών. Και αυτό δεν συμβαίνει σήμερα. Σε γενικές γραμμές λοιπόν Έχουμε στείλει τι απόψει μας. Νομίζω πως είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Είμαστε επιφυλακτικοί ε, ως προς κάποια ζητήματα. Και όπως σας είπα πρέπει να, να αναφέρουμε κάποια το τι συμβαίνει στον κόσμο σήμερα. Ευχαριστώ κύριο Σκουντής. Sorry, uh, Robert, yeah. Ήθελα να απαντήσω συντομία σε κάτι που είπε Όλε και παρεξήγησε ε, ένα νεύμα που έκανα. Φαίνεται ότι με παρατηρεί συνέχεια όλε. Δεν γλιτώνω λεπτό. Φυσικά συμφωνώ μαζί σου όλε ότι αυτά που συμβαίνουν στη Μεσογειακή Λεκάνη αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικά και καλό είναι να αναλυθούν εμβριθώς. Αλλά δεν νομίζω ότι έχουν θέση ε, σε μια τέτοια έκθεση, γιατί αυτά είναι θέματα επικαιρότητα και πολύ, πολύ γρήγορα θα μας ξεπεράσουν τα γεγονότα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη γιατί από δική μου δυσκολία δεν μπορώ να περπατήσω καλά αυτές τις μέρες. Δεν μπόρεσα να έρθω από την αρχή και να ακούσω την προφορική παρουσίαση της εισηγήτριας που όπως πάντα ξεκινάει με καλές προθέσεις κατά την άποψή μου. Το αποτέλεσμα όπως έχουμε κρίνει τουλάχιστον το διάμεσο δεν μας ικανοποίησε αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε την προσπάθεια που γίνεται. Δεν ξέρω αν συνηθίζετε κύριε Πρόεδρε επιτρέψτε μου στην αρχή να μεταφέρω δύο-τρεις σκέψεις που μου ζήτησε ο συνάδελφος ο κύριος Ντε ο Ολλανδός Ευρωβουλευτής, ο οποίος δεν μπορούσε να ήταν σήμερα εδώ επειδή έχουν εκλογές. Σύντομα λοιπόν ο κύριος De θέλει να σας εκφράσω, να σας μεταφέρω ότι ευχαριστεί την κυρία Μπερέζ για τη δουλειά που έκανε. <clears throat> Έχει δύο βασικές σκέψεις σε πολύ γενικές γραμμές, σας τις μεταφέρω. Η πρώτη είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτό που πρέπει να μας απασχολεί στην Ευρώπη είναι ένα καλύτερο και δικαιότερο σύστημα, μια ισορροπία μεταξύ πειθαρχία και κοινωνικών πολιτικών και κατά την άποψή του δεν πρέπει να διαφορούμε για τις κοινωνικές συνέπειες που έχουν αυτές οι πολιτικές και επομένως στις προτάσεις μας να περιλαμβάνεται μια ρήτρα κοινωνική, μια ρήτρα για την αντιμετώπιση της απασχόλησης. Και το δεύτερο σημείο του κυρίου Ντεγιόγκ που σας μεταφέρω σύντομα είναι ότι εν ώψη και των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου θα πρέπει να γίνει μια δημοκρατική συζήτηση και να υπάρχει μια δημοκρατική νομιμοποίηση αυτών των αποφάσεων όπου να επιτραπεί η δυνατότητα να εκφραστούν όλες οι απόψεις και να εξεταστούν με τη δέουσα σοβαρότητα ακόμα και την πιθανότητα μιας προσωρινής εξόδου από την Ευρωζώνη ενός κράτους μέλους αυτή την δυνατότητα ο κύριος Ντεγιόγκ θα ήθελε να την συζητήσουμε ή να κατοχυρωθεί εν πάση περιπτώσει στη συζήτηση και ότι εν πάση περιπτώσει να ακουστεί η γνώμη των Ευρωπαίων πολιτών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτέ είναι οι γενικέ γραμμέ οι σκέψη του κυρίου Ντεγιόγκ. Σα τη μεταφέρω με παρακάλεση διότι δεν μπόρεσε να είναι εδώ. Λίγα λόγια και από μένα τώρα σχετικά με το, το σχέδιο της τελικής έκθεσης που έχουμε. Η γενική μου παρατήρηση είναι εφόσον δεσμευθήκαμε ή έτσι το κατάλαβα, φυσικά δεν συμφώνησα, ότι το πλαίσιο της ενδιάμεσης έκθεσης δεν πρέπει να παραβιαστεί, είναι φανερό ότι σημεία με τα οποία δεν συμφωνούσαμε δεν έχουν φυγεί και επομένως δεν απαντούν κατά την άποψή μου στα προβλήματα και στις αιτίες της κρίσης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στην επικαιροποίηση που επιχειρεί με φιλότιμη προσπάθεια η συγγήτρια και με την αίρεση ότι πιθανόν να αδικώ την άποψή της επειδή είναι σύντομα γραμμένο, είναι ένα σχέδιο, τα σχόλιά μου είναι τα εξής. Πρώτον, σε σχέση με την εισαγωγή ή αν θέλετε με τη γενική αντίληψη. Δεν συμφωνώ να χωρίζουμε και να διαχωρίζουμε την κρίση της Ευρωζώνης από το ευρώ αυτό καθεαυτό. Κατά την άποψή μας εδώ υπάρχει πρόβλημα με το ευρώ αυτό καθεαυτό. Διότι έτσι όπως έχει δομηθεί και άδικα και ελλειπτικά και παράλογα ορισμένε φορές είναι φανερό ότι δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε από την κρίση της Ευρωζώνης. Άλλωστε δεν, δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω γιατί είναι παράλογα, άδικα και αναποτελεσματικά οικοδομημένο το ευρώ διότι θα σας έλεγα ότι χρειάζεται ένα κοινό νόμισμα, χρειάζεται έναν κοινό ισχυρό προϋπολογισμό και χρειάζεται και μηχανισμό δανεισμού τελευταίας καταφυγής. Εν πάση περιπτώσει χρειάζεται να καλύπτει τα κράτη με πολιτικές τις οποίες είχαν όταν είχαν το δικό τους νόμισμα και τώρα με το ενιαίο νόμισμα δεν εξασφαλίζονται. Και αυτή είναι μια βασική διαπίστωση. Επομένως δεν έχουμε κρίση της Ευρωζώνης απλά από τη μια μεριά και το ευρώ από την άλλη όλα καλώ, αν αυτό εννοεί η συγγήτρια, αλλά υπάρχει αν υπάρχει τέτοια άποψη, δεν συμφωνώ. Η δική μου άποψη είναι ότι υπάρχουν και πληρώνουμε, να το πω έτσι, τα προβλήματα του ευρώ από την ίδρυσή του, έτσι όπω τοποθετήθηκε. Η δεύτερη παρατήρηση σχετικά με το χρέο. Θα σας έλεγα ότι εδώ υπάρχει ανάγκη να γίνει μια καταγραφή στα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτό που λέγεται κρίση χρέους και εκφράζεται με τα κρατικά ελλείμματα και το χρέος αυτό καθεαυτό. Τι εννοώ με αυτό. Δηλαδή πόσο από αυτό, και αρχίζω από τη δική μου τη χώρα, πόσο από αυτό το έλλειμμα που έχει σήμερα η ελληνική οικονομία οφείλεται στην ενίσχυση των τραπεζών, τα μέτρα που πάρθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, πόσα δόθηκαν σε επιχειρήσεις που κατέρευσαν και πόσα δόθηκαν σε μια σειρά άλλα πράγματα, εμείς τα ονομάζουμε σκάνδαλα, υπερτιμολογήσεις προμηθειών, κυρίως με γερμανικές εταιρείες. Δεν λέω πως αυτή είναι η βασική αιτία. Ήδη διατυπώνεται μια, ένα αίτημα να γίνει μια επιτροπή, διεθνή Επιτροπή Λογιστικού Έλεγχου, εν πάση περιπτώσει να καταλάβουμε ποιο δημιούργησε και για ποιο λόγο το χρέο. Και βέβαια δεν θα επαναλάβω το ίδιο, την ίδια παρατήρηση, να το πω έτσι με μια απλή έκφραση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έκοψε το βήχα Δηλαδή δεν έκοψε την ισχύ και την κερδοσκοπική τάση που επέδειξαν οι οίκοι αξιολόγηση. Δεν θέλω να σα κουράζω ακόμα περισσότερο. Μια δεύτερη παρατήρηση, αν είμαι στο δεύτερο. Εντάξει, καλέ αυτέ οι σκέψει για τα ευρωομόλογα και ενδεχομένω ένα Υπουργείο Οικονομικών τη ΟΝΕ, αλλά η άποψή μου είναι ότι δεν λύνουν αυτές, αυτοί καθεαυτοί οι θεσμοί, οι νέοι θεσμοί, το πρόβλημα. Μπορεί να έχει Υπουργό Οικονομικών, δεν ξέρω τι τέτοιο, αλλά δεν θα λύσει το πρόβλημα. Είναι μια ας μου επιτρέψετε την ε, έκφραση, μια μεταφυσική αντίληψη. Εδώ πρέπει να αλλάξουν ή να μην αλλάξουν ή να τροποποιηθούν οι πολιτικές αυτές που θα υλοποιεί ο νέος, ο καινούριο, ο υπάρχον ή μη υπάρχον υπουργό οικονομικών. Εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνει αυτό, ποια πολιτική θα υλοποιεί. Ε, δεν θέλω να σας κουράσω παρακάτω ε, ε, στοιχεία. για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τα έχουμε πει πολλές φορές. Η δική μου η εμπειρία, η εμπειρία μας είναι ότι το μόνο που προσφέρει στην παγκόσμια οικονομία είναι ότι παρεμβαίνει σε περιπτώσεις οικονομικών και κοινωνικών καταστροφών και τις επιδεινώνει έτσι περαιτέρω. Επομένως, αν είναι να κάνουμε αναφορά για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λυπάμαι πρέπει να είναι αρνητικές σε κάθε περίπτωση, έτσι θα το τοποθετούσα εγώ. Τέλος, υπάρχουν και άλλες παρατηρήσεις, θα μετέχουμε στη συζήτηση, δεν θέλω να τα εξαντλήσω. Τα θέματα, μια τελευταία παρατήρηση, γενική και αυτή. Νομίζω ότι επαναλαμβάνεται ή τουλάχιστον αν το κείμενό μας θέλει να πει αυτό που τώρα θα σας πω και που επαναλαμβάνεται στα κείμενα της Κομισιόν κτλ. Ότι η στρατηγική 2020, η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης μπορεί να κατοχυρωθεί με δημοσιονομική προσαρμογή χωρίς να θυχτεί η ανάπτυξη, νομίζω ότι είμαστε στον αέρα. Δεν μπορεί να γίνει. αυτό είναι το δικό μου Δημοσιονομική προσαρμογή με, χωρίς να υπονομεύει την ανάπτυξη, το θεωρώ ασύμβατο, το θεωρώ αδύνατο. Παράδειγμα θα σας πω και θα τελειώσω. Τι ανάπτυξη να κάνει τώρα η Ελλάδα ή ενδεχομένω η Ιρλανδία. Η Ελλάδα που σε αυτή την ακραία μορφή δημοσιονομικής προσαρμογής περικόπτονται συνεχώς οι, ε, τα προγράμματα επενδύσεων. Δεν έχει καμιά δυνατότητα, κανένα μέσο ανάπτυξη. Μόνο από τον ουρανό μπορεί να προκύψει ανάπτυξη, κατά αυτή την έννοια. Επομένως αυτή τη διατύπωση τη θεωρώ ο, ασύμβατη, καθόλου πραγματική. Είναι ένας εφημισμός, δηλαδή προσπαθεί να ισορροπήσει δύο πράγματα που δεν ισορροπούν κατά την άποψη. Ε, θα σταματήσω εδώ κύριε Πρόεδρε, ενδεχομένω έφαγα περισσότερο χρόνο για την πρώτη συζήτηση και θα συνεχίσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή, την εισηγήτρια για τη δουλειά που έχει κάνει. Συμφωνήσαμε βέβαια να μην πάμε στην προηγούμενη έκθεση για το πώς θα μοιράσουμε βεβαίως τις νομοθετικές πρωτοβουλίες με τις άλλες επιτροπές και το πώς θα γίνει αυτό. Και συμφωνήσαμε και είπαμε πως θα είμαστε πολύ φιλόδοξοι. Ε, το θέμα είναι λοιπόν πώς, πώς θα τα βρούμε αυτά τα ζητήματα και να συμφωνήσουμε στο μέτρο του δυνατού. Εμείς δεν είμαστε υπέρ του να συνεχίσουμε να αναλύουμε και ζητώ συγγνώμη εδώ από τους συναδέλφους την ιστορία και την κατάσταση αλλά να πάμε παρακάτω θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια μόνο ζητήματα ένα ζήτημα που θα ήθελα να αναφέρω Εγώ θεωρώ πως θα πρέπει να αναφέρουμε το ζήτημα του δημοσίου χρέους ε, πιο συχνά. Και αυτή είναι η πρόκληση. Πώς θα, βάλουμε, πώς θα βρούμε τα προαπαιτόμενα ε, για την ανάπτυξη. Δεν, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τις αυξήσεις ε, ελλημάτων και χρέους. Αυτό σημαίνει πως θα βαλουμε πως θα βρουμε τα προαπαιτομενα για την αναπτυξη δεν μπορουμε να δούμε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο τη μέθοδο εκείνη που πρώτον θα μειώνει δραστικά το επίπεδο χρέους και ταυτόχρονα θα ε, φροντίζει την κοινωνική δικαιοσύνη και τις επενδύσεις για το μέλλον. Δηλαδή εκπαίδευση, στρατηγικές καινοτομίες, ε, ταμεία επιχειρηματικού κινδύνου για νέες εταιρείε και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ελπίζουμε να βρούμε κάποια έτσι, διατύπωση εδώ πέρα μετά. Όταν μιλάμε για τις παγκόσμιες ανισορροπίες και την παγκόσμια διακυβέρνηση. Δυστυχώς δεν συμφωνώ τόσο πολύ με ε, τις απόψεις εδώ πέρα για τη συγχώνευση των χρηματιστηρίων ε, του Euronext και τα λοιπά ε, και το αν είναι σοβαρό πρόβλημα. Αυτό είναι ζήτημα αγοράς. Δεν ξέρω αν είναι καλό για τους καταναλωτές ε, αν θα γίνουν ε, φτηνότερες οι πατάτες εάν έχουμε περισσότερες αγορές ε, στο City. Εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικό το ρόλο εδώ πέρα. Δεν νομίζω να είναι παράδειγμα αυτών των προβλημάτων. Μετά, όταν μιλάμε για το νέο νομισματικό σύστημα, για το παγκόσμιο σύστημα, πρέπει να το δούμε έτσι λίγο πιο στενά το τι πρέπει να γίνει με το δούνο του να μην είναι αποτελεί τόσο πολύ έτσι αν θέλετε ένα μαντρόσκυλο για τα κράτη-μέλη αλλά να αποτελέσει μια ομπρέλα σταθερότητας ε, κτλ. Και θα ήθελα να δούμε σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο ταυτόχρονα τα ζητήματα της χρηματοδότησης, δηλαδή το δονοτού, μετά τους πόρους, ε, το φορέας δηλαδή του περιβάλλοντος ε, και τα λοιπά, τα ζητήματα της πραγματικής οικονομίας και τα άλλα ζητήματα παγκόσμιας διακυβέρνησης. Και πράγματι η ΠΟΕ, Διεθνής Οργανισμός Εργασίας ε, και οι λοιποί που θα πρέπει να εμπλακούν πολύ περισσότερο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Τώρα δεν ξέρω αν έχει πολύ νόημα να μιλήσουμε για τους G20. Είναι μια συμμαχία με ένα είδος λέσχης. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει έτσι επίσημες τις δομές του. Αλλά που θα θέλαμε να δούμε περισσότερες συνεισφορές ε, είναι το θέμα της εσωτερικής αγοράς βεβαίως. χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ευρωπαϊκή πόρη απασχόληση, στρατηγικές ε, ε, επενδύσεων για την κοινή αγορά ενέργειας. Εκεί πέρα χρειαζόμαστε τα επόμενα βήματα και βεβαίως ε, για το Σύμφωνο Ανάπτυξης. Το δημόσιο είναι σοβαρό. Αλλά ουσιαστικό για την Ευρώπη είναι το πώς θα βρούμε χρήματα για τις πρωτοβουλίες ανάπτυξης στον ευρωπαϊκό προπολογισμό και στο εθνικό επίπεδο. Εμεί θα θέλαμε βέβαια στο το σύμφωνο ανάπτυξης. Μετά τα μεγάλα ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε. Εντάξει, κάθε ομάδα έχει τις πολιτικές της απόψεις, αλλά αφορούν για μας τα ομόλογα χρέους και τα ομόλογα έργων. Εκεί θέλουμε εμείς να αναφερθεί κάτι και βεβαίως για τον φόρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ε, είμαστε, είμαστε ε, υπέρ ε, στην ομάδα μας και θα θέλαμε να γίνει κάτι τέτοιο. You please. Joo, kiitoksia. Puhun, puhun suomea, koska täällä on erinomaisia tulkkeja. Η κυρία Γιακονσάρη, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μεταλληθώ την ευκαιρία να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Λοιπόν, έξι σημεία, αυτή είναι η διάρθρωση, πολύ ωραία. Ίσως θα έπρεπε λίγο να δούμε το ζήτημα του τι άλλαξε μετά την κρίση. Η αλλαγή είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να φανεί και στο έγγραφο, πως τα πολιτικά συστήματα κέρδισαν σε σημασία, γιατί πριν από λίγα χρόνια είχαμε αυτή την φιλελεύθερη διδαχή, αλλά τώρα θέλουμε βοήθεια από την πολιτική, η οποία πρέπει να λειτουργήσει. Αλλά τι σημαίνει αυτό συγκεκριμένα. Δεν ξέρουμε τι θα φέρει το μέλλον όσον αφορά τις μεγάλες προτάσεις της Κομισιόν για τις οποίες γίνονται διαπραγματεύσεις και εδώ μέσα γιατί βεβαίως ε, τα εθνικά κοινοβουλία θα τοποθετηθούν και δεν μπορούμε τώρα να προβλέψουμε ποιες προτάσεις τελικά θα εφαρμοστούν και θα μεταφραστούν σε πολιτικές αποφάσεις. Οπότε αυτό το οποίο δεν άλλαξε, όπως είπε και ο πρόεδρος Κλίντς, πολλές φορές είναι το ηθικό επίπεδο. Εκεί πέρα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι επικεφαλείς τραπεζίτες εξακολουθούν να έχουν τα λανθασμένα κίνητρα, θέλετε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα τελικά για να αλλάξει η ηθική, γιατί Ξακολουθούν να δρουν ε, όπως ε, έκαναν και πριν. Γι' αυτό θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για την στρατηγική της εκπαίδευσης. Ίσως θα έπρεπε να τονίσουμε αυτή την ηθική πτυχή. Εντάξει, εδώ πέρα λέμε πως ε, θα πρέπει να μπορούμε να δράσουμε. Δεν υπάρχει παραπομπή στα μπόνους λοιπά, Αλλά μιλάτε για μια στρατηγική εκπαίδευση. Δεν ξέρω, ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη γερμανική λέξη εδώ πέρα, την... που αντιστοιχεί στην παιδεία θα λέγαμε στα ελληνικά, που περιέχει δηλαδή και την πτυχή της ηθικής. για να εφαρμοστεί ε, και στην οικονομία. Ίσως λοιπόν αυτή η ηθική πτυχή ε, θα έπρεπε να τονιστεί στο κομμάτι ε, στρατηγική της εκπαίδευσης. Γιατί τελικά για την παιδεία μιλάμε. Αλλά αλλιώς η κατανομή σε αυτά τα έξι κεφάλαια είναι πάρα πολύ καλή και ελπίζω πράγματι να παραμείνουν τα κεφάλαια τόσο σύντομα γιατί αλλιώς δεν είναι και τόσο κέρια. Η Ελίζα Φερέρα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σε χαρώ την εισηγήτρια, όπως και οι προλαλήσαντες, γιατί είναι πολύ δύσκολο κατά τη γνώμη μου να συνοψίσουμε μέσα σε έξι θέματα όλα όσα είπαμε στη διάρκεια της μακροχρόνιας περίοδου ανάλυση προβληματισμού, ανταλλαγής απόψεων κτλ. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποιες πτυχές αυτών των έξι ζητημάτων και να δώσω έμφαση ορισμένα από αυτά τα θέματα. Συμφωνώ με τις έξι βασικές ερωτήσεις. Και όταν βλέπουμε το βαθμό ανάπτυξης των ζητημάτων αυτών, διαπιστώνουμε ότι ίσως πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση στο σημείο 1 που μιλάει για τις ανισορροπίες και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ζώνη ευρώ αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικώ. Σε σχέση με το σημείο 2 και 3 που είναι μεν σημαντικά αλλά εκεί γνωρίζουμε ότι η πρόοδος θα είναι πολύ πιο αργή. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε τα σημεία 1, 2 και 3, βλέπω ότι το 1 δεν είναι τόσο ισχυρό ή τόσο ανεπτυγμένο όσο θα περιμέναμε, δεδομένου ότι είναι ένα εσωτερικό πρόβλημα και πολύ σοβαρό πρόβλημα της, εσωτερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σημείο 1 λοιπόν θα πρέπει να το αναπτύξουμε περαιτέρω. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο το 1 θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τα προβλήματα του σημείου 2, δηλαδή την συνολική ανισορροπία που χαρακτηρίζει τις Ηνωμένε Πολιτείες απέναντι στην Κίνα. Δεν είναι αυτό δικό μας πρόβλημα. Εμείς έχουμε ε, στη ζώνη ευρώ σχετικά εξορροπημένο ισολογισμό. Και εξωτερική διάσταση αρκετά ισορροπημένη. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουν ορισμένες χώρες οφείλονται σε εσωτερικές ανισορροπίες της ζώνης ευρώ. Εμείς δεν έχουμε εξωτερικές ανισορροπίες, αλλά εσωτερικές. Και αν θέλουμε να κάνουμε πιο εύρωστο το ευρώ, αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το ευρώ δεν έχει τα προβλήματα που έχει το δολάριο. Η ευρωπαϊκή οικονομία δεν έχει τα προβλήματα τη αμερικανική οικονομία. Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει εσωτερικά προβλήματα και εσωτερικέ ανισορροπίε που καθιστούν πιο έθραυστο το ευρώ. Από αυτή την άποψη η πραγματική σύγκληση, η απόκληση των οικονομιών ε, δημιουργεί προβλήματα στη βιωσιμότητα των, ε, του ευρώ. Και αν θέλουμε να καταστήσουμε πιο το πιο ρωμαλαίο το ευρώ, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην πραγματική σύγκληση των οικονομιών, όχι στην ονομαστική του σύγκληση, που είναι το μόνο που μας έχει απασχολήσει μέχρι στιγμής δυστυχώς. Πιστεύω λοιπόν ότι υπό αυτή τη σκοπιά θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα και να βαθύνουμε περισσότερο στην πρώτη ερώτηση, στο πρώτο ζήτημα. Επίσης, ε, μια και θέλουμε και μια πιο μέσο και μακροπρόθεσμη προοπτική, θα πρέπει να πούμε ότι η βραχυπρόθεσμη διόρθωση των ανισορροπιών είναι σημαντική, αλλά θα πρέπει να την επιχειρήσουμε με πρίσμα μακροπρόθεσμο. Δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κοντόφθαλμα τα προβλήματα μόνο με χρονικό ορίζοντα την επόμενη διετία, αλλά να έχουμε και μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Μόνο έτσι θα είναι πραγματική η διόρθωση Αλλιώς θα μιλούμε μόνο για βραχυπρόθεσμες προσαρμογές που δεν θα έχουν βιώσιμο χαρακτήρα. Θα πρέπει λοιπόν τους στόχους μας του βραχυπρόθεσμου, να τους συνδυάσουμε με τους μέσο και μακροπρόθεσμου, γιατί μας ενδιαφέρει και η βιωσιμότητα, η διάρκεια αυτών των στόχων, ιδιαίτερα για τη ζώνη ευρώ. Μια άλλη πτυχή επίση είναι πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου. Κάτι που έχει συζητηθεί ήδη και που αφορά την εναρμόνιση τουλάχιστον της, βάσης, ε, φορολογικής βάσης του, της φορολογίας επιχειρήσεων. Μία ευρωζώνη και ένα νέο νόμισμα δεν μπορούν να λειτουργήσουν αν δεν υπάρχει μια ελάχιστη φορολογική εναρμόνιση μεταξύ των χωρών. Φυσικά δεν πρόκειται να έχουμε μια απόλυτη σύγκληση, αλλά τουλάχιστον μια συνεργασία, ένα συντονισμό στα φορολογικά ζητήματα. Για να μην είμαστε στο Κοινοβούλιο λιγότερο φιλόδοξοι από ότι οι συζητήσεις που γίνονται αλλού για το πακέτο ανταγωνιστικότητας, για παράδειγμα. Και που ούτως ή άλλως εκεί αναλύεται και αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε εμείς να μείνουμε πίσω. Ένα άλλο σημείο που δεν ξέρω αν έχει θέση εδώ ή όχι στο έγγραφο ή σε ποιο κεφάλαιο θα πρέπει να περιληφθεί είναι το, το σημαντικό ζήτημα της δημιουργίας κάποιων δομών χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Γιατί βρίσκονται ακόμη στα σπάργανα αυτές οι δομές χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή διάσταση και την εξουσία της αρμοδιότητας αυτών των αρχών. γιατί έχουμε κρίση και στις τράπεζες, αλλά και σε περίπτωση συστημικών κρίσεων, χρειαζόμαστε τέτοιες εποπτικές αρχές. Θα πρέπει να προωθήσουμε λοιπόν και αυτό το σημείο και καλό θα ήταν να το στο σημείο 1. Στο δεύτερο σημείο, συμφωνώ με τον Όλε Σμιτ. Να προσθέσουμε δηλαδή κάτι για τη σχέση μας με την παγκόσμια ανισορροπία, με τις, παγκο... τις ανισορροπίες παγκοσμίω μάλλον. Αναφέρεται ακροθυγός, αλλά καλό θα ήταν να συνδυάσουμε την μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αναπτυξιακή της πολιτική. Γιατί δεν έχει νόημα α, ε, να διαχωρίσουμε αυτές τις πολιτικές. Κάποιος που μεταναστεύει είναι πολλές φορές γιατί δεν έχει στον ήλιο μοίρα στην πατρίδα του. Θα πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε την εξωτερική μας πολιτική, την αναπτυξιακή, και έχει νόημα γιατί υπάρχουν ε, μεγάλες ανισορροπίες παγκοσμίω που πολλές φορές οδηγούν σε μετανάστευση. Επίσης γίνεται λόγος για ένα διεθνές νομισματικό σύστημα. Νόμιζα ότι ήταν ευρωπαϊκό αυτό το σύστημα που προτείνεται, αλλά βλέπω ότι θέλετε διεθνές. Θα πρέπει να γίνει μια διευκρίνηση εδώ. να μην ξεχνούμε και τη δέσμευσή μας για την πάταξη των φορολογικών παραδείσων. Το θέμα αυτό απασχολεί και τους G20. Και είναι ένα θέμα κοινό σε όλους τους υπόλοιπους στόχους, αλλά φαίνεται εξαφανίστηκε από το πρόγραμμα εργασιών μας, ενώ ίδιος ο Σαρκοζή το είχε αναφέρει. Νομίζω ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της πάταξης των φορολογικών παραδείσων θα πρέπει να είναι πολύ σημαντικός χρειαζόμαστε και μία διεθνή κανονιστική σύγκληση σε ό,τι αφορά τις χρηματαγορές. Γιατί μέχρι στιγμής ε, αναφέρεται το θέμα στον διατλαντικό διάλογο, αλλά καλό θα ήταν να γίνει το επίκεντρο αυτού του νέου νομισματικού συστήματος. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει μόνο μια αναθεώρηση των θεσμών, αλλά και των πρακτικών επιθεώρησης και των, και των κανονιστικών συστημάτων. Θα πρέπει να γίνει ένα συνδυασμό αυτών των στοιχείων. Στο σημείο 4. Καλό θα ήταν να δώσουμε περισσότερη έμφαση στην ανάγκη βιομηχανικής πολιτικής της Ένωσης και ένα σαφές οικονομικό εξωτερικό πρόγραμμα, γιατί δεν έχουμε ένα εξωτερικό οικονομικό πρόβλημα, πρόγραμμα συγγνώμη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά ήταν τα βασικά στοιχεία. Θα υποβάλω φυσικά και γραπτός παρατηρήσει μου. Γενικώ συμφωνώ με την εισηγήτρια. Τα σχόλια μου απλώ υπογραμμίζουν το ένα ή το άλλο σημείο προκειμένου να το αναδείξουν περισσότερο. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ. Πριν δώσω τον λόγο στην Περβάνς, θέλω και εγώ να κάνω κάποια σχόλια. Πρώτα απ' όλα, Περβάνς, για Νομίζω πως ε, τήρησε αυτά τα οποία είχαμε πει, δηλαδή έξι ερωτήσεις και τηρήθηκε αυτό στη δομή, οπότε διαπιστώνω πως πράγματι έτσι έγινε. Και ορθώς. Λοιπόν, η συζήτηση Η συζήτηση εστιάζεται στο ότι πρέπει να έχουμε μια σύντομη έκθεση με ξεκάθαρες ακριβείς διατυπώσεις και μια σύνοψη των προτάσεων που έχουμε. Αυτό προβλέπεται νομίζω στα συμπεράσματα. Ποια είναι λοιπόν τα συμπεράσματα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, Και αυτό έχουμε πει και στους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Πριν περάσω τώρα στα συγκεκριμένα σημεία, άλλη μια παρατήρηση για αυτό το οποίο είπε ο Λεσμίτ για τη Βόρεια Αφρική. Το θέμα δεν είναι μόνο η ανθρώπινη τραγωδία που εκτιλήσεται εκεί. Είναι και αυτό σημαντικό. Και η απέτηση για μια ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική ε, οπωσδήποτε υπογραμμίζεται. Αλλά το θέμα είναι πως ακόμη μία φορά η Ευρώπη δείχνει στην κρίση αυτή πως δεν μπορεί να δράσει. Ο ΙΕ και η ΕΠΑ αποφάσισαν ήδη κυρώσεις και εμείς ακόμα συζητάμε χαρακτηριστική συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις κρίσεις. Οικονομική κρίση, παγκόσμια πείνα, Βόρεια Αφρική. Βλέπουμε πως δεν μπορούμε να δράσουμε. Γι' αυτό είναι θέμα για εμάς, γιατί είναι χαρακτηριστικό του που πάσχουμε. Αυτό πρέπει να δούμε λοιπόν. Πρέπει να απευθύνουμε έκκληση η Ευρώπη να είναι ικανή να δράσει ως Ευρώπη. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να το πούμε αυτό στην διαμισή να μιλάει με μία φωνή, να κινητοποιείται γρήγορα, να έχει έναν εκπρόσωπο. Οπότε κάπου αυτό το οποίο είπε ο Λεσμίτ νομίζω πως είναι σημαντικό για το τι πρέπει να αλλάξει στην Ευρώπη. Για το σημείο 1, λατινικό 1, στην εισαγωγή, η κρίση, κατά την άποψή μου, εδώ πέρα δεν συμφωνώ πλήρως με τον Νικόλαο, η κρίση της Ευρωζώνης δεν οφείλεται κυρίως, δεν είναι κυρίως κρίση του ευρώ και ε, των νομισμάτων. Είναι κυρίως θέμα δημόσιου χρέους, ιδιωτικού χρέους και βεβαίως το, η έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Η έλλειψη ανταγωνιστικότητας αναφέρεται, δημόσιο και ιδιωτικό χρέος δεν αναφέρεται, εγώ θεωρώ πως θα έπρεπε να μπουν. Για το σημείο 2 Είμαστε νομοθετική επιτροπή και εδώ πέρα η Περβάνς έχει δίκιο όταν λέει πως ε, όλα αυτά που συμβαίνουν και συζητούνται στην Επιτροπή Οικονομικών δεν χρειάζεται να τα πούμε. Εμείς πρέπει να κοιτάμε μέσω μακροπρόθεσμα. Οπότε αντιλαμβάνομαι πως ε, όταν ε, πως μιλάμε έτσι για Ευρωπαϊκό Υπουργείο Οικονομικών μέσω μακροπρόθεσμα αλλά τι εννοούμε εδώ πέρα ζητήσαμε μια ενδιάμεση έκθεση και βγάλαμε τα συμπεράσματα πως μια ενιαία πολιτική, μια πολιτική για το ενιαίο νόμισμα θα πρέπει να οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερη σύγκληση των ε, φορολογικών και δημοσιονομικών πολιτικών και ίσως το Υπουργείο Οικονομικών αυτό να αποτελέσει ένα όχημα αλλά πρέπει να το καθορίσουμε σημεία 2 και 3 από την πλευρά την τυπική. Μιλάμε για παγκόσμιε ανισορροπίε και παγκόσμια διακυβέρνηση. Για την παγκόσμια διακυβέρνηση εκεί πέρα ανήκουν οι G20. Γι' αυτό νομίζω πω όλο το ζήτημα G20 που είναι στο σημείο 3 πρέπει να πάει στο σημείο 2 νομίζω. Και το Δουνουτού πρέπει να πάει συγκεκριμένα στο σημείο 3 που λέει για το νέο νομισματικό σύστημα. Όσον αφορά τώρα τις ε, συνομιλίες περί συγχώνευσης, ε, αυτό δεν τα έχουν ακόμα εγκρίνει εποπτικές αρχές για την Deutsche Börse και το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Euronext. Δεν είναι μεμονωμένο και το χρηματιστήριο του Λονδίνου συζητάει με τον Καναδά, Συγκαπούρη με Αυστραλία, δηλαδή προσπαθούν τα χρηματιστήρια μέσω συγχωνεύσεων να ενισχύσουν τη θέση τους. Γιατί, γιατί ε, χάνουν μεγάλο ποσοστό της αγοράς. Υπάρχει, ε, υπάρχουν πολλές πράξεις που γίνονται εκτός των παραδοσιακών χρηματιστηριών. Γίνονται εντός του τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή αν δείτε τις συναλλαγές των ε, γερμανικών ε, χρηματιστηρίων σήμερα είναι μικρότερο ποσοστό της αγοράς από ό,τι πριν από πέντε χρόνια. Εξού και αυτές οι συζητήσεις. Εγώ προσωπικά θεωρώ πως εάν επιτύχει αυτή η συγχώνευση υπάρχει ε, η πιθανότητα ακόμα και αν είναι αντίστροφη εξαγορά που δεν το ξέρει κανείς γιατί ούτω ή άλλω μεγάλο κομμάτι των μετόχων του γερμανικού χρηματιστηρίου είναι Αμερικανοί και αντίστροφη εξαγορά να είναι, έχουμε την ευκαιρία στην Ευρώπη να έχουμε ξανά το Euronext και την Frankfurt έτσι μαζί. Γι' αυτό νομίζω θα μπορούσαμε ε, εκεί έχετε μια προειδοποίηση. Εντάξει, αυτό είναι θετικό. Τώρα, για τις αλλαγές που λέτε. Δεν ξέρω αν χρειάζεται συμβούλιο, οικονομικό συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ. Κοιτάξτε, μην ξεχνάτε πως ο ΟΗΕ εδώ πέρα δεν ε, είναι τελείως ε, ουδέτερος. Ξέρετε πως υπάρχουν πάρα πολλά λάθη και στις εκθέσεις τους και στα Οπότε ο συνδυασμός ε, G20 και ο ΟΗΕ εγώ δεν θεωρώ πως είναι κάτι το υποχρεωτικό. Εγώ θα έλεγα πως οι G20 θα πρέπει να μετεξελιχθούν σε ένα βήμα το οποίο είναι κάτι παραπάνω από μία λέσχη συζητήσεων. Δηλαδή θα πρέπει να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα οι αποφάσεις. Αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάνουν μεγάλες ανακοινώσεις, τι θα κάνουμε κτλ. Και ε, τα τηρεί, ξέρω εγώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, λίγο η Αμερική και οι υπόλοιποι Κίνα, Βραζιλία, Ινδία κτλ. λένε καλά, κάντε ό,τι θέλετε. Εντάξει, λέμε εμεί το θα επιθυμούσαμε. Αυτή την αλλαγή πράγματι θα την επιθυμούσαμε. Τώρα για το σημείο 4, για το περισσότερο Μάριο Μόντι, ναι, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Για την στρατηγική τώρα τη εκπαίδευση. Πρέπει να λύσουμε κάτι το δύσκολο. Ξέρετε, η εκπαίδευση εξακολουθεί να παραμένει αρμοδιότητα των κρατών μελών. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε λίγο πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες οθήσεις από πλευράς Ευρώπης που θα είναι εντός των αρμοδιοτήτων όπως έχουν κατανεμηθεί αυτή τη στιγμή. Και η σκέψη δηλαδή πως χρειαζόμαστε έναν ηθικό κώδικα εδώ πέρα που ανέφερε η κυρία Γεγενσάρη είναι, είναι θετική και Πρέπει να την υποστηρίξουμε. Τώρα, για τα σημεία 5 και 6, από πλευράς λογικής, νομίζω πως το σημείο 5 που λέει πέρα από την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, να το δούμε ως πολύ μακροπρόθεσμο και άρα να πάει στο τέλος της έκθεσης. Το 6 θα το φέρνα μπροστά εγώ και το 5 τελευταίο. Από πλευράς λογικής, γιατί κοιτάει στο μέλλον. Για ε, το 6 θα ήθελα να πω το εξής. Υπάρχουν ενδείξεις, ε, καθώς ε, ερευνούν και τα κράτη-μέλη την κρίση, πως ε, τα διαρθρωτικά ταμεία δεν χρησιμοποιούνται όπως θα έπρεπε να έχουν χρησιμοποιηθεί. Δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα ανάλογα με το στόχο τους. Γι' αυτό θεωρώ πως χρησιμοποιήθηκαν τι, για, για να μπαλώσουν τους προπολογισμού όχι για να βελτιώσουν τις υποδομές των χωρών. Οπότε πρέπει να το πούμε νομίζω αυτό για να πούμε πως θα πρέπει να υπάρχει μια πιο αυστηρή επιτήρηση για να διορθωθεί αυτό στο, στο μέλλον. Αυτά από μένα. Αλλά νομίζω πως ε, μάθαμε από τη δύσκολη δουλειά της ενδιάμεσης έκθεσης. Νομίζω πως είναι πιο ξεκάθαρα τώρα τα πράγματα. Οπωσδήποτε υπάρχουν ακόμα διαφορές και βεβαίως ε, θα απογοητεύσω λίγο τον κύριο Χουντή γιατί ξέρω πως ε, και, τον κύριο Ντεγιόγκ ξέρω πως έχουν ιδέες που δεν, δεν υπάρχουν στην, στην έκθεση γιατί δεν βρίσκουν πλειοψηφίες. Αλλά νομίζω πως πρέπει να αναγνωρίσουμε πως ε, συμμετέχει, λέει τη γνώμη του και ε, συνεισφέρει σε αντίθεση με πολλούς άλλους που, που συμμετέχουν μόνο με χαρτιά. Ζαν Πολ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είχα σκοπό αρχικά να παρέμβω γιατί λόγω άλλων υποχρεώσεων ε, δεν μπόρεσα να είμαι από την αρχή στις εργασίες της Επιτροπής ε, για την αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά ακριβώς επειδή ήμουν ε, στην Επιτροπή Νομισματικών Υποθέσεων πρέπει να πω ότι συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε προηγουμένως ότι η Επιτροπή μας εδώ δεν ε, ε, είναι νομοθετική αλλά όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να προτείνει πράγματα και επομένως νομίζω ότι είναι σημαντικό να κάνει μια κρίση για τον τρόπο με τον οποίο έχουν εφαρμοστεί τα ληφθέντα νομοθετικά μέτρα. Αναφέρομαι κυρίως στην εποπτεία. Η Ελίζα ανέφερε ότι θα πρέπει να αναφέρουμε την ε, ε, εποπτεία των τραπεζών, αλλά οι αρχές ε, υπάρχουν, οι κανόνες υφίστανται. Και αυτό που με απασχολεί πολύ εμένα είναι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζομαι αυτές τις αρχές και αυτούς τους κανόνες μέσα από την ε, ε, ανάληψη καθηκόντων, από τον διορισμό ανθρώπων οι οποίοι τελικά ε, δεν έχουν την ικανότητα να ασκήσουν την εποπτεία ως θα όφυλαν. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα με τις κυβερνήσεις, με τα κράτη. Ξέρω πώς ε, εκλέγονται τα εποπτικά σώματα. Ξέρω πώς γίνονται οι διορισμοί. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν και οι επιτροπές που δημιουργούνται είναι απίστευτες. Αυτοί που δεν ε, κέρδισαν στις ε, διαπραγματεύσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και εκεί που επιτύχαμε εμείς ε, ε, σημαντικές, ε, σημαντικά στοιχεία όσον αφορά την εποπτεία, τελικά ξεπεραστήκαμε από αυτούς οι οποίοι τελικά διόρισαν ανθρώπους οι οποίοι απογύμνωσαν από κάθε νόημα την εποπτεία και νομίζω ότι το ζήτημα δεν θα πρέπει να είναι ε, εάν θα επικυρώσουμε ή όχι τους διορισμούς αυτούς, αλλά ε, στις επόμενες μέρες να δείξουμε ότι η νομοθεσία θα πρέπει να εφαρμοστεί και μάλιστα να καταδείξουμε τον δρόμο, την κατεύθυνση την οποία θα πρέπει να ακολουθήσει αυτή η νομοθεσία και ενδεχομένω έτσι δεν θα λυθούν όλα τα προβλήματα και δεν θα απαντηθούν όλα τα ερωτήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον ο ρόλο τη Επιτροπής μα εδώ ε, να ορίσουμε ε, κάποιου προσανατολισμού προσανατολισμούς ε, και να κάνουμε κάποιε προτάσει, αυτό ο ρόλο τουλάχιστον θα έχει καλυφθεί και εν πάση περιπτώσει ε, θα πρέπει να φανεί ότι η Ευρώπη προτείνει κάτι στην πλειοψηφία της ε, και απέναντι σε μια τάση επανεθνικισμού, σε μια τάση ευρωσκεπτικισμού θα πρέπει εμείς να καθορίσουμε κάποιες γραμμές, ε, κάποιες γραμμές ελπίδας για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Ζαμπόλ αν ναι, ναι, ναι, αναφέρει σύνδεση του Ζαν Πολ, θα μπορούσες να αναφέρεις πω το Κοινοβούλιο δεν είναι ικανοποιημένο με τον τρόπο με τον οποίο το Συμβούλιο, παραδιάζοντας το πνεύμα τη συνθήκης της Λισαβόνας, προχωρά διακυβερνητικά και σε σημαντικές αποφάσεις, σημαντικές και για τους πολίτες και αποφάσεις με κόστος όταν μιλάμε για τη μόνιμο ταμείο διάσωση, αφήνει απ' έξω το κοινοβούλιο. Δεν είναι σωστό αυτό. Και πρέπει να, να το πούμε. Κάτι τελευταίο για την έκθεση. Είπα πως απάντησαν 15 κράτη-μέλη στο, στο ερωτηματολόγιο. Κοιτάξτε, δεν, είναι, δεν πρόξενη η έκπληξη το ότι είναι πολύ, πολύ επιφυλακτικά τα Εθνικά Κοινοβούλια για περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη Ευρώπη, περισσότερο προπολογισμό κτλ. Είναι πολύ επιφυλακτική γιατί ε, δεν ξέρω, ίσως να μην έχουν ασχοληθεί πολύ με το θέμα, αλλά εν μέρη φοβούνται ε, πως θα χάσουν επιρροή. Όπως και να έχουν τα πράγματα, θα πρέπει να τους ε, πείσουμε και βέβαια αυτό θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Ε, γι' αυτό όμως ακριβώς θεωρώ πως πρέπει να αναφερθούν αυτά τα σημεία. Και κάτι ακόμα για την έκθεση. Πρέπει να είναι σύντομη, ευανάγνωστη, όπως είπε ο Ζαμπόλ, και είναι σε καλό δρόμο η ως προς αυτό. Αλλά στο τέλος, όταν έχουν τελειώσει όλες οι ψηφοφορίες, να θέλουμε να τεκμηριώσουμε την εργασία που έχει γίνει εδώ πέρα. Έχουμε πολλές εκθέσεις, ε, ε, εργαστήρια, ακροάσεις, όλα αυτά θα πρέπει νομίζω να πάνε σε έναν τόμο. Όπως υπέβαλαν οι Γάλλοι φίλοι νομίζω, για να φανεί ακριβώς το, να καταγραφεί το έργο της Επιτροπής και τώρα εάν θα είναι έτοιμο κάτι τέτοιο πριν το καλοκαίρι ή μετά το καλοκαίρι δεν έχει τόσο σημασία αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να περιέχει όλα τα έγγραφα, τα πρακτικά και τα λοιπά. Λοιπόν, Περβάνς, έχει το λόγο. Πολύ ωραία. Αν έχω τον χρόνο που θέλω, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλους. Ε, γιατί είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε και τον χρόνο μέχρι τώρα να κάνουμε έτσι μια πολύ σε βάθος ε, ανάλυση. Ε, χρόνο έχουμε βέβαια, βλέπω ότι κάποιοι συνάδελφοι έχουν φύγει, εν πάση περιπτώσει. Πρώτα απ' όλα, σημειώνω ότι υπό την αίρεση της δικής σας προτάσεως κύριε Πρόεδρε ε, να αντιστρέψουμε τα σημεία 5 και 6 που ε, πραγματικά θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα και την δέχομαι. Ε, διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση εδώ της διαδομής της έκθεσης. Από την μία πλευρά λοιπόν συμφωνώ το 5 να γίνει 6 και αντίστοιχα να επαναοργανώσουμε επίσης τα σημεία 2-3 ε, και συμφωνώ απολύτως γιατί εδώ άλλωστε έχουμε απέναντί μας μόνο το προσχέδιο άρα αυτού του είδους οι διαφορετικές κινήσεις ε, θα γίνουν και επίσης ασχολούμαι αμέσως με αυτό που είπε ο συνάδελφος Όλη Σμιτ που θα πρέπει να αποτελέσει και ε, κατά κάποιο τρόπο που αφορά και την εισαγωγή και το σημείο 6. Συμφωνώ με αυτά που είπε. Έστω και αν μιλάμε για την οικονομική, χρηματοπιστωτική, κοινωνική κρίση, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε πλήρως μία αναταραχή η οποία μας αφορά άμεσα εμάς σαν Ευρωπαίους γειτόνους. Και θα ήθελα να πω τρία πράγματα για την έκθεσή μας. Βλέποντα για τη γλώσσα του σώματος ε, των συναδέλφων. Πρώτον, τα όσα συμβαίνουν στην Αφρική μας υπενθυμίζουν ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε την αξία των ε, θεμελιωδών μας αξιών, της δημοκρατίας δηλαδή, της ε, προσδοκίας ε, προς την πρόοδο βάσει της εκπαίδευσης και βεβαίως την ισότητα. Δεν τα ξεχνάμε αυτά και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Ένα δεύτερο σημαντικό μήνυμα το οποίο φωτίζεται και από την ιστορία ε, και άλλωστε ο Σμιτ ε, είπε προηγουμένως ότι το μέλλον έρχεται από το παρελθόν. Πρέπει να πω το εξής. Ε. Εξεπλάγει όταν έπεσε ο Μπεναλή. Γιατί είδα ένα παραλυσμό με αυτά που είχαν συμβεί όταν άλλαξε καθεστώς η Ουγγαρία. Τότε θυμάμαι ότι ήμουνα υπεύθυνη ε, βοηθός του Λορόν Φαμπιούς, υπεύθυνη για τέτοια θέματα. Και είχα αναλάβει την οργάνωση μιας, ε, ε, ενός συνεδρίου που είχε τίτλο «Άνοιγμα προς, προς την Ανατολή, κίνδυνοι και προσδοκίες» και ευκαιρίες μάλλον. Αυτό είναι ένα διώνυμο το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Από τη μία μεριά οι κίνδυνοι και από την άλλη μεριά οι ευκαιρίες. Ε, τι να σας πω, ενδεχομένως δεν μαθαίνουμε ποτέ από τα παθήματα του παρελθόντος, έστω και αν το προσπαθούμε. Ε, και βεβαίως ξέρουμε ότι οι τράπεζες μας είναι έτοιμες να δώσουν λεφτά στις χώρες αυτές αλλά γιατί βεβαίως το χρήμα είναι εύκολο και ξέρουν ότι θα τους φέρει πολύ χρήμα αλλά υπάρχουν άλλα ζητήματα τα οποία είναι πιο σημαντικά. Είναι η εκπαίδευση, είναι η οικοδόμηση ενός κράτους δικαίου, ε, είναι η ε, ανοικοδόμηση βάσει της ισότητας και της δημοκρατίας έτσι ώστε να αποφευχθούν τα φαινόμενα ε, διαφθοράς. Αυτά θα έπρεπε να είναι τα πιο σημαντικά πράγματα έτσι ώστε να οικοδομηθούν σύγχρονα κράτη με σωστή αστυνομία, με δικαστικές αρχές, ε, με ε, δημοσιονομικές φορολογικές αρχές οι οποίες θα μπορούν, θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν το κράτος να λειτουργήσει δημοκρατικά. Και το τρίτο είναι αυτό το οποίο αναφέρατε άλλωστε, ε, όπως και στη διάσκεψη της Κομπεχάγης τι να σας πω τώρα, μπορώ να κάνω λίγο δημαγωγία γαλλική, πρέπει να πω ότι α, η κυρία Άστον δεν είπε και τίποτα καλύτερο από αυτά που είπε η κυρία Λιώμαρη, η δικιά μας η Γαλλίδα υπουργό. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν είναι το ουσιώδες εκεί. Το ουσιώδες είναι ότι είναι οι γειτονές μας, ε, είναι δικιά μας ε, ε, πολιτική ευθύνη, ιστορική ευθύνη. Και εδώ βλέπουμε ότι σε αυτή την κρίση φαίνεται ότι τα πρώτα μηνύματα τα στέλνουν οι ΗΠΑ. Εν πάση περιπτώσει. αυτή τη στιγμή εγώ εκφράζω την επιθυμία το μήνυμά μας να είναι σαφές, ευανάγνωστο και συνοπτικό. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Σημείωσα όλες τις παρατηρήσεις της κυρίας Μπαστός. Όμως, δεν θα συμφωνήσω απολύτως μαζί της. Στο, το κείμενο το οποίο έχετε εδώ μπροστά σας είναι αποτέλεσμα της ε, εργασίας της γραμματείας επί τη βάση των υποδείξεων των πολιτικών ομάδων. Αυτό είναι το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε. Και εάν δεν θεωρείτε το κείμενο αυτό είναι το σωστό αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, τότε δεν ξέρω πώς να τι μπορεί να αποτελέσει βάση εργασίας. Και πρέπει να πω επισήμως ότι για μία ακόμα φορά αυτό το πόνημα είναι εργασία της, Επιτροπ... της ε, Γραμματείας που βασίστηκε στα όσα είπαν οι πολιτικές ομάδες. Βεβαίως δεν υπάρχουν όλα αυτά που είπε ο καθένας, γιατί πρέπει να γίνονται και κάποιες επιλογές. Και αυτό που πρέπει να κάνω εγώ σαν εισηγήτρια είναι βασιζόμενη σε αυτό το κείμενο το γραπτό και στη σημερινή μας συζήτηση να περάσω ένα σαφές ευρωπαϊκό πολιτικό μήνυμα. 28 euh, euh, και από αυτή την άποψη θα ήθελα να αναφέρω ότι σχετικά με τις εργασίες με το κείμενο του ΕΛΚ έχω μια δυσκολία. Το πρώτο έγγραφο το οποίο μου δόθηκε λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επικεντρωθεί στις κύριες δραστηριότητες της, άνω και κάτω τελεία, υπηρεσίες. Δεν συμφωνώ όμως και το λέω σαφώς. δεν νομίζω ότι συζητήθηκε πολύ το ζήτημα αυτό πριν γραφτεί έτσι. Γιατί η επικέντρωση στις υπηρεσίες για να παραχθεί τη θέμενη αξία <laughs> μα ήδη η κρίση μας οδήγησε σε τελείως διαφορετικά συμπεράσματα. Ε, Δηλαδή ότι χρειαζόμαστε τη βιομηχανία, χρειαζόμαστε ε, τις υπηρεσίες, αλλά χρειαζόμαστε και τη γεωργία, χρειαζόμαστε και ε, ε, την, ασφάλεια, χρειαζόμαστε την διατροφική ασφάλεια. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να συμφωνήσω με την πρόταση έτσι όπως έχει γραφτεί σε αυτό το κείμενο, αλλά μπορώ να συζητήσω με ε, το ΕΛΚΑ. Μπορούμε να συζητήσουμε να δούμε. Ε, τώρα νομίζω ότι η συνένεση είναι σαφής πάνω σε πολλά σημεία. Στα υπόλοιπα σημεία με την κυρία Μπάστο συμφωνούμε. Όλοι Σμιτ, σας ευχαριστώ για τα όσα αναφέρατε. Νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Όταν συνδέεται την οικονομική πραγματικότητα με την ε, μετανάστευση, σε έναν ιδεώδη κόσμο λέτε ότι θα πρέπει να ανοίξουμε την αγορά στα προϊόντα τους, στα προϊόντα των χωρών αυτών και όχι στους μετανάστες τους. Ναι, εντάξει, αλλά μην ξεχνάτε ότι εμείς έχουμε και δημογραφικό έλλειμμα και ότι, όπως είχε πει και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών πολύ παλιότερα εδώ, η Ευρώπη θα χρειαστεί ε, τα εργατικά χέρια της Αφρικής. Ε, τα χρειαζόμαστε ήδη σήμερα και θα τα χρειαζόμαστε και αύριο. Αλλά αυτό που θα αλλάξει μετά από όσα συνέβησαν στην Αφρική είναι ότι σε αυτές τις χώρες θα υπάρξει ένα άλλο οικονομικό μοντέλο. Και επομένως θα επιστρέψουν, όπως συνέβη και στην Ισπανία παλιότερα και στην Πορτογαλία, θα επιστρέψουν πολλοί μετανάστες στις ε, χώρες τους, στις χώρες προέλευσής τους. και προτείνω να ε, πούμε κάτι γι' αυτό και νομίζω ότι για τους μετανάστες και για την καλύτερη ένταξή τους στα νομικά μας συστήματα στις χώρες μας θα πρέπει να προβλέψουμε πραγματική ισότητα δικαίου για τους μετανάστες όσους μείνουν εδώ και όσους θα εξακολουθούν να δουλεύουν εδώ. Τώρα, τι να σας πω, ε, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρατε μετά είναι σημαντικά. Η αξιολόγηση των ε, δαπανών, των εθνικών ε, δαπανών γίνεται και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα σε μακροοικονομικά πλαίσια και νομίζω ότι ενισχύεται με τον τρόπο αυτό η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Χουντή, Αυτά που λέτε για την κοινωνική ρήτρα βεβαίω, το γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα συμμερίζομαι απολύτω. Και επίσης ε, θα σας δικαιώσω και για ένα άλλο σημείο. Όταν λέτε δηλαδή, μετά από αυτά που είπε ο κύριος Σμιτ, ότι βεβαίως βρισκόμαστε σε κρίση της Ευρωζώνης και όχι του Ευρώ. Όλη αυτή η κρίση, και το έχουμε πει και το ξαναπούμε, δεν αμφισβητεί κανείς αυτή την κρίση το ίδιο το ευρώ. Ε, ναι, εντάξει, ο κύριος Βιλάν στη Γαλλία έλεγε ότι είναι ερετικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ακούγονται διάφορες φωνές, αλλά ε, στην ουσία δεν αμφισβητεί κανείς ε, ότι πρέπει να υπεραμεινθούμε του ευρώ. και είδαμε ότι όταν και οι πολιτικοί βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, όταν στριμώχνονται, παίρνουν κάποια μέτρα τα οποία βασίζονται και στο ευρώ και θέλουν να στηρίξουν το ευρώ. Ε, και βεβαίως μπορεί να ε, και, και παίρνουν θέσεις ε, ε, οι οποίες τελικά ε, σώζουν το ευρώ και η καγκελάριος Μέρκελ και ο πρόεδρος ε, και ο διοικητής της τράπεζας ο κύριος Τρισέ πήραν τελικά τις αποφάσεις που έπρεπε. Αλλά είναι γεγονός ότι το Μάστριχτ έχει ξεπεραστεί πλέον. Πέρασαν χρόνια από την θέση σε ισχύ του ευρώ. Και με την κρίση αυτή την οποία διανύουμε υποχρεώμαστε να λάβουμε υπόψη αυτό που λέει η κυρία Φερέιρα. Δηλαδή, οι ε, εσωτερικές ε, ισορροπίες έχουν γίνει πιο σοβαρές από τις ε, εξωτερικές ανισορροπίες. Εξού και το ερώτημα το οποίο θα συζητήσουμε με τον Ζακ Ντελόρ στις 14 Μαρτίου που θα μας τιμήσει με την παρουσία του. Τι γίνεται και πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Βεβαίως μπορεί κανείς να παίξει με τα ε, λόγια ε, και να πει ότι δεν αμφισβητείται το νόμισμα. Ε, ναι, εντάξει, αμφισβητείται η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ωραία, αυτή τίθεται να αμφιβόλω. Με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επιτύχει και όχι μονάχα σε χρηματοπιστωτικό επίπεδο και εκεί συμφωνώ με τις ανησυχίες του κυρίου Χουντή. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Βλέπω τι γίνεται στο Συμβούλιο. Εγώ όμως θα ήθελα να συμφωνήσουμε εδώ μεταξύ μα για να πούμε ότι η πραγματική διαθροτική μεταρρύθμιση την οποία χρειάζεται παντού η Ευρώπη είναι το ζήτημα της εκπαίδευσης. Αυτή είναι η πραγματική διαθροτική ε, μεταρρύθμιση. Πρέπει να δούμε πώς θα την κάνουμε και πώς θα τη χρηματοδοτήσουμε. Ευχαριστώ την κυρία Πιτικάνεν για την στήριξή της και βεβαίως ε, έφυγε. Ε, αυτό ε, το διόνυμο το οποίο και εκείνη ανέφερε, δηλαδή ε, χρέος κρατών και ανάπτυξη. Όσον αφορά το χρηματιστήριο, και επανέρχομαι εδώ σε αυτά που είπε ο πρόεδρος, βεβαίως καταλαβαίνω ότι η Deutsche Börse θέλει να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της αλλά εμείς σαν νομοθέτες θα πρέπει να δούμε τι επιπτώσεις έχει η όποια κίνηση κάνει και ποια, και, και είναι η δυναμική που δημιουργείται. Και ειλικρινά σας λέω, θα ήθελα να έχω μια σαφή εικόνα ε, του, του τι σημαίνει Deutsche Börse. Δηλαδή ποιοι έχουν κεφάλαια, τα κεφάλαια του χρηματιστηρίου. Στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή, στην έκθεση Σουιμπέρν, είχα κάνει μία τροπολογία ε, στην οποία διαπίστωνα ότι το, ε, το πνεύμα της ε, ΜΥΦ τελικά είχε εντελώς αλλάξει από την παρουσία της Ντάρπουλ. Και αυτό ήταν σημαντικό. Δεν έγινε δεκτή η τροπολογία. Αλλά εγώ συμφωνώ μαζί σας, συμμερίζομαι την ανησυχία σας για τη λειτουργία της Ντάρπουλ. Δηλαδή τι θα γίνει, οι νομοθέτες πρέπει να επιβάλλουν, να υποχρεώσουν την αγορά ε, να έχει διαφάνεια. Και το γεγονός ότι ε, τα χρηματιστήρια είναι θύματα ας πούμε, της λειτουργίας του Ντάρπουλ δεν δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Και ε, επίσης υπάρχουν και πολλές επενδυτικές μεγάλες τράπεζες, οι οποίες δεν είναι καν ευρωπαϊκές. Και ξέρετε, είχαμε πάει μαζί στις Ηνωμένε Πολιτείε και το είχαμε ε, και το θέμα των αντισταθμίσεων ο στόχος των επενδυτικών Αμερικανικών τραπεζών είναι να έχουν μονάχα αντιστάσματα στην Νέα Υόρκη. Ε, και εγώ πιστεύω ότι ε, αυτή η συγχώνευση τελικά σε αυτό το στόχο αποσκοπεί. Μπες με θα τα ξανασυζητήσουμε. Θα επανέλθω ε, σε αυτά που είπε... Bildung, parce que... ναι, ναι, η γνώση μου της ε, γερμανικής δεν είναι τόσο καλή ώστε να καταλάβω το κείμενο στο οποίο αναφερθήκατε. Θα με βοηθήσει ο Ζαμπολ κοζέ. Ε, στην συνάδελφο Φερέιρα, ε, ναι, βεβαίως το ζήτημα της πραγματικής σύγκλησης ή ονομαστικής σύγκλησης είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Ε, επίσης, όπως είπα και προηγουμένως, το θέμα της μετανάστευσης για μένα είναι θέμα ισότητας και ε, ισότητας δικαίου. Ναι, δεν αναφέραμε τους ε, φορολογικούς παράδεισους στην αρχή, αλλά γιατί το έκανα γιατί το, το ζήτημα αυτό και στο ΖΕ20 μάλλον θα περάσει έτσι χωρίς να συζητηθεί και πολύ. Στον Πρόεδρο απήντησα και για τη συγχώνευση και για το Συμβούλιο, α, για το ε, Συμβούλιο Οικονομικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών. Τι να σας πω, ίσως δεν το δουλέψαμε πολύ το θέμα αυτό, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια ε, συνάντηση με τους ε, για να δούμε τι θέλουμε να βάλουμε στο κομμάτι αυτό. Κοιτάξτε, αν έπρεπε να είχα οργανώσει μια ομάδα εργασίας ε, για την διακυβέρνηση, εγώ θα την είχα κάνει ε, τελείως διαφορετική. Ήταν ο κύριος Σενζόν. Τέλος πάντων, ε, ε, ήταν ένα σωρό άνθρωποι, αλλά τελικά τα συμπεράσματά τους δεν, ήταν, δεν έβρισκαν σύμφωνους όλους. Ας προσπαθήσουμε εμείς τουλάχιστον να πάμε λίγο πιο πέρα, γιατί το είπαμε και στην πρώτη έκθεση ενα z G20 το οποίο είναι τόσο δεν είναι καθόλου συγκεκριμένο και απλώς ακροθυγός ε, αναφέρει κάποια πράγματα, ε, επιτρέπει και στους Κινέζους ε, να μην είναι ε, να, να μην είναι απολύτως ε, κατά. Ε, επίσης ένα νομισματικό ταμείο, διεθνές νομισματικό ταμείο έτσι όπως είναι τώρα επιτρέπει σε πολλούς να ξεφεύγουν και να μην αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα προβλήματα με συγκεκριμένο και ουσιώδη τρόπο. Επομένως κάτι πρέπει να γίνει και σε αυτό. Κύριε Γκοζές, σας καλώ να διαβάσετε το 5-3 αυτού του προσχεδίου που ετοίμασε η Γραμματεία, γιατί είναι ακριβώς αυτό που ε, αναφέρατε και πιστεύω ότι το, στην έκθεση αυτή θα πρέπει πραγματικά να γίνει ε, αναφορά ειλικρινής στην άποψη που έχουμε για την, ε, τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει η χώρα η εποπτεία αυτή τη στιγμή και πώς εφαρμόζονται οι κανόνες της ε, εποπτείας. Και οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και οι πόροι έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε... Ε, να έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη αλλά και μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης των αρχών αυτών. Τελευταία παρατήρηση είναι τεχνικής φύσεως. Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι τελικά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τις εργασίες της ε, Επιτροπής μας. Και γνωρίζοντας τι συμβαίνει στις ε, Επιτροπές Έρευνας του Γαλλικού Κοινοβουλίου, <laughs> θα ήθελα εδώ να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να καταλήξουμε κάτι, ε, κάπου. Αλλά να μην αποσιωπήσουμε την σημασία και την ποιότητα της εργασίας του, των εργασιών που κάναμε στο πρώτο τμήμα, στην πρώτη φάση. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να διασυνδέσουμε τις δύο φάσεις και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να μείνουμε πιστοί ε, και στο σύνολο των ε, συμβολών που έκαναν οι διάφοροι συνάδελφοι και όλοι αυτοί με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή στην διάρκεια της πρώτης φάσης. Ευχαριστώ πολύ τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την έντονη συζήτηση και τη συμμετοχή. Καλημέρα σας εύχομαι. Ευχαριστώ.